Um, okay, colleagues, I think we can make a start. I apologize for starting a bit late, but I... Να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Λυπάμαι λοιπόν, που καθυστέρησα. Talking about public... με είχαν ε, σε μια συνέντευξη και μιλούσα για τις δημόσιες προμήθειες, καταλαβαίνετε. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην τελική μας τελευταία συνεδρίαση πριν από τις θερμινές διακοπές. Θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο θέμα σήμερα το οποίο θα μας, μας πάρει τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα να το ολοκληρώσουμε. Μία γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού για το κοινωτικό σήμα και η νομοθεσία των κρατών μελών που έχουν να κάνουν με το κοινωτικό σήμα. Αυτά φυσικά είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά για την λειτουργία της ιστορικής αγοράς και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι η αρμόδια για το πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα, τα γενετικά δικαιώματα, αλλά όλοι φυσικά έχουμε συναρμοδιότητα και μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν ε, την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης, μπάστο, ε, κυρία Στάιλερ. Είσαστε σκιώδης για το θέμα αυτό. Θέλετε να είστε σκιώδης ε, για το θέμα αυτό σήμερα το απόγευμα. Είναι και τα γενέθλιά σας. Όχι, όχι, γενέθλια έχω στα τέλη του μήνα, πρόεδρε, και στις 4 θα πρέπει να είμαι στην Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Και θα είμαι εδώ μέχρι τότε. Κύριος Παντσέρη, κύριος Κρόιτσμαν, κυρία Ρούλε. Νομίζω ότι η κυρία Ρούλε κάνει πιο πολύ τη σκιώδη ηγήτρια από ότι και εγώ. Και εγώ θα είμαι σκιώδη, φαντάζομαι, από τη δική μου ομάδα. Έχουμε λοιπόν του συνήθει ύποπτου σήμερα το απόγευμα. Από την Επιτροπή έχουμε τον αρμόδιο για, από τη Γενική Διεύθυνση Πνευματικών Δικαιωμάτων. Θα σας δώσουμε το λόγο και από το Αλικάντα, από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς. Έχουμε έναν εκπρόσωπο. Έχω επισκεφθεί το Αλικάντα και ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη η επίσκεψη και η κυρία Μπάστος ασφαλώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάστος καταρχάς και μετά να ακούσουμε ίσως κατευθείαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει μερικά στοιχεία και μετά να ακούσουμε και τους κοιόδης. Νομίζω ότι καλά θα τα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, μια σκηνή πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σα δίνω το λόγο λοιπόν, κυρία Μπάστο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρωτογαλλικά. Σας ευχαριστώ πάντω για την παρουσίαση αυτή τη έκθεση προσπαθήσω να πλαισιώσω αυτές τις δύο εκθέσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού και της οδηγίας για το κοινοτικό ε, σήμα μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με βάση το Small Business Act του 2008 και την ε, οδηγία περί διανοητικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν σε έναν διτό στόχο. Καταρχήν να ανταποκριθούμε στη συνθήκη της Λισαβόνας και να θίξουμε αυτό το κοινό θέμα ως προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Το δεύτερο στόχο θέλουμε να διευκολύνουμε την ζωή των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ και των καταναλωτών ως προς την βελτίωση, τον εξορθολογισμό και τον εξυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η κατάθεση του κοινοτικού σήματος και μείωση των δαπανών και των ε, πολυσχηδών διαδικασιών, έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές να γίνουν ταχύτερες, πιο προβλέψιμες και με μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συνενετικό πλαίσιο, δηλαδή ότι το κοινοτικό σήμα εντάσσεται στον θεμητό ανταγωνισμό και σχετίζεται με την ε, προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η διάκριση των προϊόντων και των αγαθών, καθώς και των υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν καλύτερα τους πελάτες τους ή επιχειρήσεις. Μέσα από τα σήματα υπάρχει μεγάλο δυναμικό καινοτομίας. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η σωστή ένταξη του κοινοτικού σήματος στο νομοθετικό μας έργο και αυτό ευεργετεί βεβαίως και την απασχόληση. Αυτή η πιο σύγχρονη νομοθεσία που εισαγάγουμε με την αναθεώρηση αυτή θα προωθήσει την επένδυση, τις επενδύσεις, θα δημιουργήσει νέα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες και θα υποβοηθήσει και τους καταναλωτές μέσα στα πλαίσια της ζωτικής σημασίας προστασίας τους και δημιουργία νέας απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιμέρους εθνικά ε, σήματα τα οποία εναρμονίστηκαν εδώ και 20 χρόνια και το κοινοτικό σήμα θεσπίστηκε εδώ και 15 χρόνια. Και πρόσφατα διενεργήθηκε μία μελέτη από το Ινστιτούτο Max Planck για την πνευματική ιδιοκτησία. Μπορώ να σας πω ε, επί παραδείγματι ότι το 2012 ε, είχαμε 75.900 αιτήσει για σήμα σε αντίθεση με τις 40.000 ορισμένων ετών πριν. Αυτό το νέο σύστημα κοινοτικού σήματος είναι ένα εύρωστο σύστημα το οποίο μας απασχολεί διαχρονικά. Το 2011 το Ινστιτούτο Εναρμόνισης του Κοινοτικού Σήματος ε, έλαβε την ε, χιλιοστή αίτηση από τη στιγμή της δημιουργίας του. Γι' αυτό είναι πολύ ε, θετική η πρόταση Επιτροπής, δηλαδή η υποβολή αυτού του πακέτου και η αναδιατύπωση της οδηγίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται μεγάλη αναδιατύπωση, διότι η, βάση, η νομική βάση ισχύει. Θέλουμε μόνο να εξυγχρονίσουμε καλύτερα αυτό το πλαίσιο για να έχουμε ένα πιο φτηνό και αποτελεσματικό σήμα. Σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα έχουμε την ευκαιρία να κατανοήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και της Επιτροπής. Θα ήθελα όμως να επισύρω την προσοχή σε ορισμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να επαναδιατυπωθούν. Λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση της νομοθεσίας και επειδή θέλουμε το σήμα να είναι πιο προσβάσιμο, ο ετών θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στον Εθνικό Οργανισμό καταρχήν, όπου θα ε, τύχει μεγαλύτερης βοήθειας, δηλαδή το Εθνικό Ινστιτούτο θα είναι ο μεσάζων έναντι του νέου οργανισμού κοινοτικού σήματος. Έτσι, θα συνεργαστούμε με τους εθνικούς οργανισμούς σε πρώτη φάση. Οι ετούντες λοιπόν θα έχουν αυτό το εθνικό εφαλτήριο. Ως προς την εκτίμηση, τη γενικότερη εκτίμηση για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ελάφρυνση του κόστους προς τα, τις ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει γενικότερη εποπτεία των επιχειρήσεων, διότι έχει μεγάλη σημασία η βοήθεια προς τις ΜΜΕ που δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα για τη συνεχή διαβούλευση των, ως προσθετήσεις αυτές. Γιατί πολλές φορές δεν υπάρχουν και αρκετοί εντολής που μπορούν να προωθήσουν αυτά τα αιτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τα σήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε σύγχυση και γι' αυτό θα πρέπει ε, ο καταναλωτής να μην οδηγηθεί σε εσφαλμένη επιλογή. Έμπρακτα λοιπόν Οι ετούντες θα πρέπει να γνωρίζουν εγκαίρως τα δικαιώματά τους. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κατά προτεραιότητα δικαιώματα, καθώς και τις επενδύσεις και το εμπλεκόμενο κόστος για την έγκριση του κοινοτικού σήματος, έτσι ώστε να μην έχουμε άσκοπα έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό καταχώρησης το οποίο να είναι ενιαίο. Μπορούμε λοιπόν να ελαφρύνουμε το συνολικό κόστος για να επιλύονται εγκαίρως και διαφορές όπου ανακύπτουν. Αυτό προβλέπεται από δύο κράτη-μέλη. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ε, μας απασχολεί είναι τα τέλη που προβλέπονται από ένα συγκεκριμένο άρθρο του, της οδηγίας. Ε, σε περίπτωση αναθεώρησης των τελών θα πρέπει να δούμε που υπάρχουν αποκλίσεις. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο οργανισμός αυτός για την ε, συνολική βελτίωση του συστήματος των σημάτων και να μην μεταφέρεται εάν υπάρχει πλεόνασμα στον γενικό προϋπολογισμό. Ως προς το Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει απόκληση στον αριθμό της σύνθεσης, δύο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να υπάρχει καλή αντιπροσωπευτικότητα έτσι ώστε να υπάρχει ισόβαθμη και ισόνομη ε, πρόσβαση. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπάρχει θεσμική εξισορρόπηση κατά την εποπτεία και τη διαχείριση του Ινστιτούτου. 5. Ε, έργο του οργανισμού. Έργο και καθήκοντα. Αυτά δεν πρέπει να ορίζονται εκ των υστέρων αλλά εκ των προτένων. Και ως προς την ανάθεση νέων καθήκοντων θεωρούμε ότι ε, όλα τα προϊόντα θα πρέπει να την χάνουν της ίδιας ε, προστασίας. Και ο ίνος ε, και τα ποτά, τη στιγμή που προέρχονται από μια συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να βρίσκονται εκτός αρμοδιοτήτων του οργανισμού. Στο άρθρο 123β1 ορίζεται αυτό. Αυτά είναι ορισμένα από τα σημεία που θέλουμε να θίξουμε με τις δύο αυτές γνωμοδοτήσεις και όπως σας είπα αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος με μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τους σκιώδεις. Είμαι πεπισμένη ότι θα βρούμε ένα κατόφλι συνεννόησης και έναν κοινό παρονομαστή. Είμαι στη διάθεσή σας και τέλος θα ήθελα να πω σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ότι δυστυχώς είμαστε μακριά από αυτό που θα επιθυμούσαμε. Το αποφάσισε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αλλά καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι γνωμοδοτήσεις να μεταφραστούν τάχιστα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου έτσι ώστε να διευρυνθεί και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Θα ήθελα να μας πει και η Προεδρία της Λιθουανίας πώς θα προωθήσει το θέμα αυτό και ποιο είναι το, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι Πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα, παρακαλώ του σκιώδεις να λάβουν και αυτοί το λόγο. Σκιονίχ, ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την ολοκληρωμένη περιγραφή της πρότασης. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, διότι η εισηγήτρια Αναφέρθηκε στα βασικά χαρακτηριστικά της δέσμης μέτρων. Το βασικό όμω χαρακτηριστικό του συστήματος προστασίας του κοινωτικού σήματος είναι ότι είναι δι της φύσης υπό την έννοια ότι τα σήματα προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο καταρχήν από τα αντίστοιχα γραφεία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και ο άλλος πυλώνας είναι το κοινωτικό βεβαίω το οποίο προστατεύεται από το γραφείο στο Αλικάντε και όπου εκεί κατατίθενται σήμερα τα οποία την χάνουν αυτομάτως κοινωτικής προστασίας σε όλη την κοινωτική επικράτεια. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, κάθε χρόνο περίπου 100.000 αιτήσει υποβάλλονται στο γραφείο του Αλικάντε και περίπου άλλες 400-500.000 αιτήσει σε εθνικό επίπεδο. Το οποίο σημαίνει ότι τα περισσότερα σήματα επιζητούν προστασία σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία να συνεχιστεί η εφαρμογή αυτού του διτού συστήματος και στο μέλλον. Δεν υφιστάται λοιπόν ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσης. Η ανάγκη είναι να εξυγχρονίσουμε να κάνουμε πιο αυτοσυνεπές το σύστημα, να προάγουμε την ενερμόνιση, διότι η χρησιμότητα των εθνικών συστημάτων δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες για κάποιο λόγο έχουν μόνο τοπικές δραστηριότητες, σε εθνικό δηλαδή επίπεδο. Πολλές επιχειρήσεις πριν καν προσφύγουν στο Αλικάντε θα αξιοποιήσουν ένα, δύο, τρία εθνικά γραφεία, μια μικρομεσαία επιχείρηση παράδειγμα που κάνει τα πρώτα βήματα. Έχει σημασία λοιπόν να είναι εναρμονισμένε οι εθνικέ νομοθεσίε για αυτού του είδου, η τη κλίμακα τη επιχειρήση. Θέλω να πω δηλαδή ότι οποιαδήποτε επιχείρηση, ότι μάλλον δεν είναι δεδομένο ότι οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία θέλει να διεθνοποιηθεί προσφυγεί κατευθείαν στο Αλικάντε. Γι' αυτό και έχει σημασία σε ένα προγενέστερο στάδιο οι εθνικέ νομοθεσίε να είναι εναρμονισμένε. Αυτό έχει σημασία και ενδιαφέρον τι επιχειρήσει. Χρειάζεται επίση να εξυγχρονίσουμε το σύστημα για να συνάδει με τι ε, ανάγκε των συγχρόνων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων και για να εξασφαλίζεται προστασία στο εθνικό και στο κοινωνικό επίπεδο. Θέλουμε να καταγράψουμε τις βέλτιστες πρακτικές που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο, ώστε αυτές οι καλές πρακτικές να διατεθούν σε όλους τους χρήστες ανά την Ευρώπη. Να δούμε δηλαδή με ποιο τρόπο εύκολα, γρήγορα και φτηνά μπορεί κάποιο να υποβάλει όχι μόνο αίτηση, αλλά να υποβάλει και ενστάσεις χωρίς να υπάρχει ανάγκη να καταφεύγουμε στα δικαστήρια. Να επιλύονται όλα αυτά δηλαδή σε διοικητικό επίπεδο. Και θέλουμε η διαδικασία στο Αλικάντε να διευκολυνθεί και αυτή, να έχουμε λιγότερε καθυστερήσει, η καταχώρηση να γίνεται το σύντομα των δυνατών και με τρόπο πιο στοχευμένο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία μεταξύ των εθνικών γραφείων σημάτων. Απαιτείται σαφή νομική βάση προς τον σκοπό αυτό και χρηματοδότηση βεβαίω για την χρηματοδότηση σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος και κοινή βάση δεδομένων μεταξύ άλλων. Κατά τα άλλα, η πρόταση προβλέπει άλλα σημαντικά στοιχεία αντιμετώπιση της απάρης, για παράδειγμα, των κλεψίδικων και καθεξής. Να πω και δύο λόγια για τα όσα ανέφερε η συγκητρία. Η δυνατότητα των ετούντων να υποβάλουν αίτηση για κοινοτικό σήμα στο εθνικό όμω γραφείο σημάτων. Αυτό δεν υπάρχει πια ως δυνατότητα. Και τούτο διότι δεν υπάρχει πρακτική, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μιλάμε για πολύ λίγε αιτήσει, διότι όλοι πηγαίνουν κατευθείαν στο Αλικάντε. Παλιά υπήρχαν δυσκολίε που δεν υφίστανται όμω πλέον. Η συγγήτρια είπε επίση ότι Τεχνικά γραφεία δεν έχουν πλέον την υποχρέωση να εξακριβώνουν κατά πόσον προϊφιστάμενα σήματα, ενδεχομένω αντιστρατεύονται το υποαίτηση σήμα. Δεν πρόκειται πλέον για υπηρεσία. Είναι απλώς εμπόδιο. Πολλέ φορέ σταματούν κάποιε αιτήσει ε, χωρί να υπάρχει λόγο. Διότι τα προηγούμενα δικαιώματα πολλέ φορέ είτε δεν αξιοποιούνται, μπορεί θα έπρεπε να διαγραφούν ουσιαστικά από τα Μητρώα, είτε οι κύριοι του δεν μπορούν καν να αντιπιστούν ε, Κάποιε επιχειρήσει εξαφανίστηκαν, δεν υπάρχουν πια, μετακινήθηκαν κ.ο.κ. Συνεπώ πιστεύουμε ότι αυτή η πρακτική αποτελούσε και θα αποτελούσε εμπόδιο και δεν πρέπει να περιπτώσει να γίνεται αντικείμενο επίκληση για την απόρριψη μια αίτηση. Όμω, οι υπηρεσίε ενημέρωση πρέπει να παρέχονται, πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε τέτοιου είδου υπηρεσίες στους χρήστες. Τέλος, το οικονομικό μέρο. εάν υπάρξουν πλεονάσματα από το ΓΕΑ, τι θα γίνει. Αυτό αποτελεί και απόδειξη ότι το κινητικό σήμα βεβαίω ε, είναι επιτυχία, αποτελεί επιτυχία. Λοιπόν, στους ε, οικονομικούς κανόνες προβλέπεται ότι δεν πρέπει να προκύπτει πλεόνασμα. Παρά το γεγονό ότι το Γραφείο Ενερμόνησης ε, έχει αναλάβει και άλλες δραστηριότητες, περιπτώσεις παράβασης. Για παράδειγμα, θα απαιτηθεί χρηματοδότηση και πλέον δραστηριότητες που θα προσθεθούν, αλλά ο στόχος τελικός είναι να υπάρχει ένα πλεονάσμα, αλλά αυτό να μεταφέρεται στον κοινοτικό προπολογισμό, το οποίο είναι λογικό. Αυτό είναι και ένα μικρό αντάλλαγμα αν θέλετε με την έννοια ότι στην περίπτωση ελλείμματος θα κληθεί ο κοινωτικός προπολογισμός να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα αυτό. Αυτά εντάχει. Περιμένουμε ενδιαφέρον την συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Να ακούσουμε και τους ε, σκιώδεις Κρότσμαν Μπίλεν και ο κύριος Έγκστρομ. Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά δεν έχουμε άλλον από τους σοσιαλιστές. Κρότσμαν πρώτα απ' όλα. Κύριε Κρότσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κοινωτικού σήματος θεωρώ ότι αποτελεί μια καλή βάση γιατί ε, εμείς γνωμοδοτούμε στην αρμόδια Επιτροπή. Πολλά στοιχεία της ε, οδηγίας ε, θεωρώ ότι είναι σωστά. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορική αγορά και τα τελευταία ζητήματα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρώτη φορά θα έχουν τη δυνατότητα τα παραποιημένα ε, προϊόντα που περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλους προορισμούς να τα κατάσχουν μέσα των τελωνίων. Και εδώ υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία. Και αυτό το επιβεβαίωσε και η απόφαση του δικαστηρίου το 2011. Τα μέτρα για τα προϊόντα τα παραποιημένα, τα οποία είναι σε διαμετακόμιση μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν περιορισμένα τώρα. Και η αφαίρεσή τους από το εμπόριο θα είναι βασικό μέσο και θα, επιτευ, επιτευχθεί αυτό με, το, τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήμουν τον Ιούνιο ε, αρμόδιος για την έκθεση για τον κανονισμό για τα πειρατικά προϊόντα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να περάσει το μέτρο να υπάρχει σωστός έλεγχος από τα τελωνία. Και με τη νέα πρόταση θα μπορούμε να αφαιρέσουμε και από το εμπόριο τα προϊόντα αυτά και η νέα νομοθεσία φαίνεται να είναι πιο απλοποιημένη γιατί τύφονται και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και βάσει της κρύψης πρέπει να υπάρχει δράση και σε περιπτώσεις διαμετακομίσεις Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί το εμπόριο με τις άλλες τρίτων με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα γενώσιμα, σε περίπτωση φυσικά που δεν υπάρχει παραβίαση της εμπορικής νομοθεσίας. Οι επιχειρήσεις δεν θα επωφεληθούν όμως από την προστασία το, της αγοράς το σύστημα που προτείνεται σε ό,τι αφορά τα τέλη θα ωφελήσει ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί θα ζητήσουν μία προστασία αγοράς που θα ταιριάζει στις ανάγκες τους και σε τέτοιες περι... Περι περιόδου κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνονται τέτοια μέτρα τα οποία θα προωθούν την αγορά, την ανάπτυξη, τι επιχειρήσει, θα μειώνουν τη γραφειοκρατία χωρίς όμως να επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους ε, προπολογισμού. Αυτά χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση για το ότι ε, εξυπηρετούν τα μέτρα αυτά και το κινητικό σήμα την ιστορική αγορά. Αλλά μετά από 20 χρόνια χρειάζεται μια ανανέωση. Ελπίζω λοιπόν η οδηγία αυτή να μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στην τρέχουσα θητεία. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Well, certainly we would... Um, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα όχι, φυσικά δεν θα θέλαμε να χάσουμε και τη δική σας τεχνογνωσία γιατί είσαστε ε, εισηγητής για τη σχετική οδηγία και νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς ε, και να συνδράμουμε στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σα είπα ότι είμαι σκιώδη και είναι ένα από τα ε, πιο αγαπημένα μου θέμα, θέματα. Και εμεί ακόμα πιστεύουμε ότι είναι καλά τα κοινωνικα θύματα. σήματα. Όταν γράφει Coca-Cola απ' έξω, ξέρω ότι είναι ευθύνη τη Coca-Cola και ξέρω επίση ε, που μπορώ να βρω άλλη μια Coca-Cola αν μου αρέσει το προϊόν. Και αυτό μα οδηγεί ε, στη δευτερεύουσα συνέπεια. Είναι καλό να υπάρχει ανταμοιβή των εταιριών αυτών. Είναι δευτερεύον, αν θέλετε, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Μα αρέσουν λοιπόν τα κοινωνικά σήματα. Και θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με κάτι που η κυρία Μπάστος και άλλοι. Έχουμε ένα καλό σύστημα κινητικού σήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1996 όταν εισήχθη, κανείς δεν ήξερε αν θα λειτουργήσει σωστά, αλλά λειτουργήσε. Άρα, εν γέννη, πρέπει να πω ότι σε περίπτωση αμφιβολίας ας αφήσουν τα πράγματα όσο έχουν, γιατί λειτουργούν σωστά και καλά. Φυσικά πάντα υπάρχει περιθώριο για μικρές βελτιώσεις. Να θυμόμαστε όμως ότι λειτουργεί καλά το κοινωτικό σήμα, τα εθνικά σήματα λειτουργούν καλά και ότι το σύστημα αποσκοπείται να τα συνδέσει καλύτερα. Για το θέμα εν προκειμένου. Πολλά από τα στοιχεία είναι λεπτομέρειες τεχνικές, τεχνικής φύσεως. Κανα δύο σημεία προφανώς θα είναι ακαθόδη Καταρχάς, όπως είπε ο κύριος ε, Κρόιτσμαν, τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή των δικαιωμάτων εμπορικού σήματος στην Ευρώπη, ώστε να καλύπτει και τις περιοχές ελεύθερου εμπορίου και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια αρκετά σημαντική αλλαγή και διεύρυνση. Τα εμπορικά σήματα πάντα είναι περιορισμένα γεωγραφικά αν θέλει κανείς ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα, εθνικό σήμα. Αυτά ισχύουν σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο αντίστοιχα. Άρα μπορεί κανείς να έχει ένα εμπορικό σήμα στην Ευρώπη, αλλά κάποιος άλλος να έχει το ίδιο σήμα στην ε, Νοτιοαμερική, στην Ασία, ούτω καθεξής. Αν το δίκαιο, λοιπόν, το ευρωπαϊκό ε, συμπεριλάβει και προϊόντα που περνούν μέσω μετακόμιση από την Ευρώπη, αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί αν είναι παραποιημένο το προϊόν το οποίο αποστέλλεται για να φτάσει στην Ευρώπη, αυτό είναι παράνομο και θα έπρεπε να θεωρείται παράνομο. Χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία, ίσω και καλύτερα μέτρα για να πιάσουμε τα προϊόντα αυτά. Αλλά να διευρύνουμε την νομοθεσία και κάποιο ο οποίο νόμιμα έχει παράγει κάτι στην Κίνα και θέλει να το στείλει στην Νότια Αμερική μέσω του Ρότερνταμ και να μην μπορεί επειδή υπάρχει το αντίστοιχο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα, θεωρώ ότι αυτό φτάνει πάρα πολύ επιζήμιο για το νόμιμο εμπόριο, για το λιμάνι του Ρότερνταμ. Και φυσικά αυτό έχει μεγάλες συνέπειες, μεγάλο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. σχόλια εκτός μικροφώνου του κ. Κρότσμαν. Θα πρέπει να μιλήσετε και στους ακτιβιστές για τα φάρμακα για το θέμα αυτό. Εγώ απλά αναφέρω τι θα σας πούν. Δεν θα χαρούν ασφαλώς. Αν σταματήσουν οι αποστολές αυτές για νόσιμων φαρμάκων στο λιμάνι του Ρότερνταμ λόγω παραβίαση τη νομοθεσία. Και προφανώ θα υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο με την νομοθεσία αυτή. Ένα άλλο ζήτημα. Όπως όλοι ξέρουμε, είχαμε και την έκθεση Κρόετσμαν για τα πνευματικά δικαιώματα και τότε το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι το σωστό που έπρεπε να γίνει είναι να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης. Αν ο έμπορος ε, μπορούσε να αποδείξει ότι υπάρχει πελάτη στην άλλη χώρα θα ήταν εντάξει. Αυτό το απέρριψε το Συμβούλιο. Ακόμα και αυτή η αρκετά ήπια δηλαδή διάταξη την απέρριψε το Συμβούλιο, την ε, άφησε να περάσει. Να το θυμόμαστε αυτό. Και τώρα βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πηγαίνει πολύ πολύ πολύ παραπέρα. Ούτε καν ε, θα αρκούσε η αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Άμεση καταστροφή του προϊόντος. Δεν νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν. Μου προκαλεί κάπως έκπληξη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έξι μήνες μόνο έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο σαφώ τη θέση του για το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αυτό που τη ζητήσαμε. Τι να πω. Κάτι άλλο αμφιλεγόμενο. Προτείνουν τα τελωνία να έχουν δικαίωμα κατάσχεσης προϊόντων που αγοράζω εγώ από έμπορο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ως ιδιώτης αγοράζω κάτι από το Hong Kong, το τελωνίο θα μπορούσε να έχει δικαίωμα να το κατάσχει, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως να είναι απόλυτα νόμιμα προϊόντα τα οποία πολλούνται νομίμως στο Χονγκ Κονγκ. Αν εγώ προσπαθήσω να τα αγοράσω, το τελωνίο έχει δικαίωμα κατάσχεσης. Με αυθαίρετο τρόπο από δική μου άποψη. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και να περάσουμε στα πιο τεχνικά ζητήματα. η έρευνα εξ που ανέφερε η κυρία Μπάστος. Στην παρούσα φάση αυτό υπάρχει σε περίπου 12 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφωνώ, αλλά διαφέρει η κατάσταση σε διάφορες χώρες. Και αυτές οι χώρες θέλουν να έχουν τη διαφορά αυτή. Εγώ δεν βλέπω γιατί αυτό θα πρέπει να εναρμονιστεί δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να το απαγορεύσουμε αυτό στην ε, Σουηδία, για παράδειγμα. Αν θέλει, να το διατηρήσει. Ε, για το κοινωτικό σύστημα, φυσικά και το κοινωτικό σήμα, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκή διαδικασία, αλλά νομίζω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν τι θέλουν. όταν ε, ε, η απάντηση είναι θετική, καταφατική ε, και υπάρχει τέτοια αυταπάγγελτη έρευνα, είναι οριστική η απάντηση. Ενώ σε άλλε περιπτώσει ίσω να μην είναι. Για τι μεγάλε επιχειρήσει, ξέρετε, αυτό δεν κάνει καμία διαφορά, γιατί έτσι κι αλλιώ έχουν δικού του εμπειρογνώμονε και δίκη τεχνογνωσία. Κάτι άλλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει, να εξαναγκάσει τα κρατη να συνεργαστούν. Εγώ δεν είμαι κατά της συνεργασίας και η δική μου εμπειρία γιατί εργαζόμουν στο σκανδιναβικό, στη σκανδιναβική υπηρεσία για τις ευρεσιτεχνίες η ανεπίσημη συνεργασία λειτουργεί πάρα πολύ καλά, αλλά ο εξαναγκασμός, αν θέλετε, σε συνεργασία των κρατών μελών, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, θεωρώ ότι δεν είναι καλή ιδέα. Να έχουμε επίση υπόψη ότι στην παρούσα φάση τα πράγματα πήγαιναν αρκετά καλά από μόνα του. Νομίζω καλό ήταν να το αποφύγουμε αυτό. Και τέλο α περάσουμε στο ψητό, στα χρήματα. Υπήρξε μεγάλο πλεόνασμα. Και αυτό, όπω λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μια ένδειξη ότι το σύστημα λειτουργεί καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όλοι θέλουν τα χρήματα αυτά και οι ε, Εθνικές Υπηρεσίες Ευρεσιτεχνίας. Δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτεί κυβερνητικές υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες που θέλουν να συντηρούν. Νομίζω ότι το πιο λογικό είναι οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύπτει να μεταφέρεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πρόκειται για ευρωπαϊκή υπηρεσία και οι πιο πολλές υπηρεσίες ε, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτή βγάζει κάποιο πλεόνασμα. Φυσικό θα ήταν να μεταφερθεί το πλεόνασμα αυτό στον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά ασφαλώ αυτό θα το συζητήσουμε επί μακρόν. Επίσης, να σας πω ότι στην Επιτροπή Γιουρή ο εισηγητής ε, ε, ήταν έκπληκτο από τον τρόπο που είναι δομημένο το πακέτο αυτό. Με οδηγία και κανονισμό, εντάξιος εδώ. Αλλά τα τέλη τα αφαιρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα επεξεργάζεται μόνη της πριν διαμορφωθεί το σύστημα για το εμπορικό σήμα. Ίσως πιο λογικό θα ήταν να αποφασίσουμε τι θα γίνει με τα διάφορα κομμάτια, τμήματα του εμπορικού σήματος και μετά να δούμε τι γίνεται με τα τέλη. Πρέπει να ομολογήσω ότι και εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την έκπληξή του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει προσαρμογή και ορισμός των τελών προτού αποφασίσουμε ποιες θα είναι αυτές οι υπηρεσίες και πώς θα διαμορφωθούν. Μάλιστα και στο σημείο αυτό θα κλείσω νομίζω. Του των λαχθέντων να σας πω ότι προσβλέπω στην μελλοντική μας συνεργασία για το θέμα αυτό. Όπως σας είπα, μια φορά έχουμε και ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί καλά. Συζητάμε να κάνουμε κανένα δυο μικρές βελτιώσεις και αλλαγές. Δεν είναι τίποτα πιεστικό. Αν είναι πολύ φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θεωρώ. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πραγματογνωμοσύνη αυτή, η οποία είναι πολύτιμη για την κυρία Μπάστος. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί καλώς. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Έγκστρομ με ακούει. Δεν νομίζω. Θα ήθελα να σχολιάσω και να σας πω ότι το ότι θεωρείται το σύστημα λειτουργεί καλώς μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι όλα είναι καλώς. Επειδή επισκέφθηκα τον οργανισμό, Μπορώ να σας πω ότι η τεχνολογία και η δυνατότητα έρευνα σε τράπεζες δεδομένων έχει αλλάξει τη διάσταση του ζητήματος, έχει αλλάξει τις διαστάσεις γενικότερα του όλου θέματος. Προσπαθούμε να μειώσουμε το χρόνο υποβολής αίτησης. Ίσως ε, έχετε απόψεις, κάποια άποψη επί του θέματος. Ο κύριος Μπίλαν. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε το λόγο. Όχι, ο κύριο Μπίλα. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο για τη συζήτηση, γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ήδη ασχοληθήκαμε με τα εμπορικά σήματα από την Επιτροπή Γιούρη. Εγώ ήμουν εισηγητής για μια τέτοια έκθεση και αυτό που έχει σημασία είναι το παρατηρητήριο κατά της παραχάραξης αγαθών. και είναι η δραστηριότητά του. Κατανοήσαμε ότι είχε μεγάλη σημασία να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις στα πλαίσια των εξελίξεων της αγοράς των παραχαραγμένων αγαθών. Κάτι το οποίο δεν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και οδηγεί σε απώλειες, σε ζημίες δημοσιονομικού ε, περιεχομένου, τα διάφορα εξαρτήματα, τα παιχνίδια, ο οικιακός εξοπλισμός, ε, σε αυτούς τους τομείς η παραχάραξη θα μπορούσε να σταθεί επιζήμια και για την ανθρώπινη ζωή γι' αυτό. Θα πρέπει να βασιστούμε στον Εθνικό Οργανισμό εμπορικού σήματος. Είδαμε ότι δεν υπάρχει συνεργασία όπως θα επιθυμούσαμε και αυτό μπορεί να, δώσει μεγαλύτερη, να προσδώσει μεγαλύτερη σημασία στη λειτουργία του οργανισμού. Θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα απολούστευσης, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, που θα οδηγήσουν στην προστασία των επιχειρήσεών μας. Γιατί πολλές επιχειρήσεις που θέλουν να καταγραφεί το εμπορικό του σήμα, θα πρέπει να κατανοήσουν, να γνωρίζουν πολλούς κανονισμούς στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να απλουστεύσουμε τα μέτρα έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για αυτές τις επιχειρήσεις. Υπάρχει, ένα, υπάρχει το κοινοτικό σήμα το οποίο αποτελεί μεγάλο ευεργέτημα για τις επιχειρήσεις, αλλά οι κανονισμοί μας θα πρέπει να είναι πιο ακριβείς, ιδιαίτερα για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί. Γι' αυτό έχει σημασία η συνεργασία και με τους εθνικούς οργανισμούς εμπορικού σήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλά σχόλια τα οποία θα χρησιμεύσουν στην κυρία Μπάστος. Να της δώσω ίσως τον λόγο για κάποια καταρρυτικά σχόλια και να δούμε και το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα. Obrigada, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, Κρόισμαν, Άγκστρονγκ και Λιπούς για, τη, για τις θετικές τους απόψεις κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής η οποία ε, σχετίζεται με τη δική μας πρόταση αναδιατύπωσης και εναρμόνισης Έχουμε ορισμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να χτενίσουμε, ιδιαίτερα ως προς τα πλεονάσματα και τους τελικούς αποδέκτες και θα ήθελα να βασιστούμε το ότι θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η εργασία εγκυρότητας, το σύστημα λειτουργεί καλώς, θα πρέπει όμως να το προσαρμόσουμε στη συνθήκη της Λισαβόνας και να βασιστούμε στους οργανισμούς, τους αποκεντρωμένους εθνικούς οργανισμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξεκινάμε εκ του μηδενός. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό κατόφλι και η ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών αποτελούν ένα μέσο για την ε, τελειοποίηση του συστήματος που είναι ένα σταθερό σύστημα. Επίσης, ο οργανισμός του Αλικάντε θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς και αρμοδιότητες που να τον καταστήσουν πιο αποδοτικό για να υπηρετεί τους εθνικούς οργανισμούς και να προστατεύει τα συμφέροντα των ΜΜΕ. Προς τα εκεί κινούμαστε και ιδιαίτερα για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Εκεί θα επικεντρωθούμε. Θεωρούμε ότι σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να έχουμε τον μέγιστο κοινό παρονομαστή για να μπορέσουμε να τελειοποιήσουμε ένα σύστημα που γενικά είναι θετικό. Έχουν συνεισφέρει πολύ και πολλαπλώς ως προς ε, πρακτικής υφής ζητήματα και επίκαιρα ζητήματα αντιμετώπισης της παραχάραξης και θα πρέπει να ανταποκριθούμε και στις διάφορες προκλήσεις έτσι ώστε να μειώσουμε το κόστος των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά, το κόστος λειτουργίας, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό είναι το σημείο εκκίνησης που μας βρίσκει σύμφωνους, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις μικρές αποκλίσεις οι οποίες είναι πρόδειλες από αυτή την πρώτη φάση ανταλλαγής απόψεων και που θα μας απασχολήσουν στο εγγύς μέλλον και μεσοπρόθεσμα. Για τα δύο αυτά ζητήματα σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. thank you very um, Φαντάζομαι θα αφιερώσετε ένα μέρο του καλοκαιριού σα στη συγγραφή τη νομοδότηση, γιατί πρέπει να είστε έτοιμοι 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθο. Καλή επιτυχία. Μετά, 25 Σεπτεμβρίου θα να πούμε για συζήτηση. 26 Σεπτεμβρίου είναι προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Όπω είπε η κυρία Δουλεύουμε σχεδόν τόσο γρήγορα όσο η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, γιατί εκεί θα πάμε 5 Νοεμβρίου, οπότε μέχρι τι 17 πρέπει να έχουμε τελειώσει με τη συζήτηση και τις τοπολογίες. Θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Κύριε βέβαια αν υπάρξουν αλλαγές θα μας ενημερώσει στο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστώ και τους παρατηρητές από το Γραφείο Νερμόνησης Εσωτερικής Αγορά. Και περάμε στο δεύτερο σημείο. Για μια βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία το 2020. Έχω τον κύριο Κοφράτη εδώ, ο είναι ο μας. Έχω τον κύριο Μπόρισοφ και δεν ξέρω αν ο κύριος Κρότσμαν θα παραστεί. Α, ναι. Ο κύριος Κρότσμαν και τον κύριο Χατζημαρκάκη. Εγώ είμαι εδώ πάντως, αυτό είναι βέβαιο, εκ μέρους της ομάδας μου. Έχουμε λοιπόν την χαρά από εδώ και πέρα. Ακούσουμε τον Και επί των 52 τροπολογιών έχω μία σύντομη συνάντηση σήμερα το απόγευμα και για αυτές, οπότε θα ψηφίσουμε τον Σεπτέμβριο. Κύριε Σιγητά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους, τους κοιόδης ιδιαίτερα, ότι τους απέστειλα χτες ένα πρώτο κείμενο προτάσεων τροπολογιών συμβιβασμού σε σχέση με τις προγενέστερες τροπολογίες που μου είχαν αποστείλει. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας ε, μέσα στα πλαίσια της σημερινής συζήτησης. Και τις δύο επόμενες ημέρες θα ήθελα να μου στείλετε τα γραπτά κείμενα με τις παρατηρήσεις σας. Διότι, όπως θύμισε και ο πρόεδρος, ε, έχουμε πολύ ε, χαμηλό περιθώριο διότι θα ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Ε, τελειώνουν οι εργασίες μας αυτή τη βδομάδα και θα ψηφίσουμε αμέσως όταν ξαναρχίσουν οι εργασίες μας το Σεπτεμβρίο. Παρά το πολύ στενό χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε μεγάλες δυσκολίες διότι η προτάσεις μου αποστήλατε εμπλουτίζουν την αρχική πρόταση και γι' αυτό δεν υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες νομίζω, αντίθετα, ότι όλα θα λειτουργήσουν ε, τάχιστα και αποδοτικά. Σε σχέση με το κείμενο που σας είχα υποβάλει, προσέθεσα μέσω των δικών μου τροπολογιών ορισμένα επιχειρήματα τα οποία για λόγους χώρου δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό κείμενο. Ιδιαίτερα ως προς τη σήμανση των καυσίμων με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και υπογράμμισα τη σημασία των επενδύσεων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την καινοτομία, ορίζοντας 2020 καθώς και θέματα οδικής ασφαλείας. που θα μπορούσε να μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες σήμερα τεχνολογίες. Οι τροπολογίες μετατράπηκαν σε συμβασμούς, όχι όλες βέβαια, και οι συμβιβασμοί αφορούν το θέμα των επενδύσεων. Ο συνάδελφος Μπόρισοφ μου έκανε υποδείξεις και μετά υπάρχει και το θέμα της αλυσίδας των προμηθετών που απασχόλησε τους Μπόρισοφ και Βέσπαλ το θέμα των ε, εξαρτημάτων, Χατζη Μαρκάκης και Μπόρισοφ μου απέστειλαν ε, σημαντικές ε, παρατηρήσεις, τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και τα χρησιμοποιημένα οχήματα, που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον ε, πρόεδρό μας. Υπάρχουν και ορισμένα επιπρόσθετα θέματα ως προς την αναδιάρθρωση της βιομηχανικής πολιτικής, ιδιαίτερα ως προς την αυτοκινητοβιομηχανία, με συναφείς ε, πολιτικούς τομείς, όπως ο τομέας της ενέργειας. Υπάρχουν και μεμονωμένες τροπολογίες που είναι θετικές και που στα συμπεράσματα θα εκτιμήσω. Μπορώ να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα. Την τροπολογία Μπόρισοφ σε σχέση με τις σχέσεις ε, με τις τοπικές αρχές για τη δημιουργία μιας αγοράς για τα ηλεκτρικά οχήματα και ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε ιδιαίτερα που μας ε, ανέφερε και ο πρόεδρος αφορά τη δική μας συμμετοχή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή και ιδιαίτερα την δική μας Επιτροπή στις εργασίες της Επιτροπής, ξεκινώντας από την εργασία του προγράμματος CARS 2020. Εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε δυνάμει της προγενέστερης εμπειρίας μας και του κειμένου, του αρχικού κειμένου και των τροπολογιών. Άρα καλυπτόμαστε από τους συμβασμούς και τις τροπολογίες όπως υποβλήθηκαν. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου αποστείλετε όχι μόνο παρατηρήσεις, αλλά και γραπτά κείμενα μέχρι την ε, Πέμπτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μία σύνοψη και χωρίς φόβο και πάθος να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Μπορώ να σας ε, ενημερώσω λέγοντας, μπορώ να σας απαντήσω μετά από την ανταλλαγή απόψεων, εν είδη συμπεράσματος. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για τη σπουδή σας να προτείνετε συμβασμούς. Ας ακούσουμε από τους σκιώδεις, ο κύριος Μπόρισοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην ε, κατάρτιση του κειμένου ως εκπρόσωπος της ομάδας του ΕΛΚ. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από την ε, έκθεση. Υπάρχουν καλές ε, ιδέες, ελπίζω να είναι καλές και συμβαστικές τροπολογίες. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε πόσο σημαντικό είναι ο κλάδος αυτός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να υπάρχει σαφή σήμανση για τον καταναλωτή. Όλα αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά καθώς ε, οδεύουμε προς το 2020 θα πρέπει να είναι και εφικτή η στόχη αυτή και άρα θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ των μέτρων και της χρηματοδότησης, ανάλογα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κινητοβιομηχανία. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω τις εξή τροπολογίες, να επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα για να είναι καλές οι εξαγωγές μας και προκειμένου να έχει πρόσβαση ο Ευρωπαίος πολίτης σε καλές τιμές και καλή ποιότητα. Αυτό με έρευνα και ανάπτυξη και Χρησιμοποιώντα όλα τα οικονομικά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά δεύτερον, για να είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να φροντίσουμε το νομικό πλαίσιο που διέπει την αυτοκινητοβιομηχανία να είναι αρκετά ευέλικτο, προκειμένου να ανταποκρίνεται γρήγορα στι νέε τεχνολογικέ αλλαγές, στι καινοτομίε, που αποτελούν και τη βάση του ανταγωνισμού τρίτον μεγάλη σημασία δίδονται στα οχήματα ιστορικής σημασία και στην νομοθεσία για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Τα οχήματα αυτά είναι τμήμα της κληρονομιάς μας, της ιστορικής μας κληρονομιάς και δεν μπορούμε να τα καταργήσουμε όπως άλλα οχήματα. Επίσης πιστεύω ότι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να υποστηρίξουν την αυτοκινητοβιομηχανία από τους χώρους στάθμευσης, από τις ε, διοικητικές διευκολύνσεις. Κοιτάξτε, κάποιες περιοχές ήδη εφαρμόζουν τέτοια μέτρα και καλό θα ήταν να βελτιωθεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι πάροχοι, γιατί είναι ο κινητήρας της καινοτομίας και παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζουν ακόμα τεράστια προβλήματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την έβρεση λύσεων που φωτεριάζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχω εννέα τροπολογίες και όπως είπε και ο κ. Κομπεράτη, όπως μαζί της θα τις καταθέσω μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Κρότσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφο Χατζημαρκάκη δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Ευχαριστεί ιδιαίτερα τον εισηγητή για την πολύ καλή δουλειά του. Ο κ. Κομπεράτη ήδη στη γνωμοδότηση του έθιξε πολλά σημαντικά ζητήματα. Οι τροπολογίες του εισηγητή αλλά και οι υπόλοιπε τροπολογίες είναι ισορροπημένες και νομίζω ότι ε, ωφέλουν το κείμενο. Ο συνάδελφος Χατζημαρκάκης θέλει να φέρει δύο θέματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκινητικότητα και κατά δεύτερον, ε, τη δημιουργία μια ενιαία ε, ευρωπαϊκή αγορά για εξαρτήματα. Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πολλά έχουν συζητηθεί, δεν υπάρχουν όμω συγκεκριμένε προτάσει. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προχωρούν πάρα πολύ αργά. Είναι ακατανόητο ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να υπάρξει ένα ενιαίο πρότυπο για μια διαπαφή. Η ανάπτυξη επίσης ε, της ε, σχετικής υποδομή είναι πολύ βασικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν εθνικές προδιαγραφές στην Ευρώπη που απαγορεύουν την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς για το tuning. Και τις, ε, θα πρέπει εδώ να, να σημειωθεί πρόοδος για να διευκολυνθεί η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αγοράς. Πρόκειται για μια αγορά όπου υπάρχει μεγάλο δυναμικό, αλλά αυτό έχει παραμεληθεί. Και στον κλάδο αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί. Ε, Εκτός μικροφώνου. Δυστυχώς, δεν λάβαμε τις επιπρόσθετες ε, τροπολογίες του εισηγητή. Να επανέλθω σε ένα θέμα, γιατί σε ό,τι αφορά την, ε, τις κρατικές επιδοτήσεις μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αυτό το ακούσαμε Μα όταν μιλάμε για την αυτοκινητοβιομηχανία η οποία τα πηγαίνει καλά, ξεκινάμε και μιλάμε για κρατικέ επιδοτήσει, η οποία τα πηγαίνει μόνη τη καλά ο κλάδο αυτό. Είναι από μόνο του αποδοτικό. Μου προκαλεί έκπληξη. Uh, well, I'm sure that you'll the amendments. Ναι. Ε, δεν είχα τους πράσινους κάποιον ε, σκιώδη για το κείμενο. Λοιπόν, δύο λόγια μόνο γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, Γιατί τη δεσμή τροπολογιών, όπως είπε και ο κύριος Κοφεράτη, ε, σίγουρα βελτίωσε το κείμενο. λίγο ησυχία παρακαλώ στην αίθουσα. Βλέπω μια πολύ καλή έκθεση. Ε, Επίση, εξαιρετικέ είναι και οι συμβαστικέ τοπολογίε. Γενικώ, ο κ. Κοφεράτη, από ό,τι φαίνεται, θα δεχθεί όλε τι άλλε τοπολογίε, Τι ε, συμβαστικέ. Ε, και το ίδιο ισχύει και για τι ε, μη συμβαστικέ. Αλλά θα τα δούμε στην ψηφορία. Παρά αύριο θα έχουμε μια απάντηση. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την έντονη να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Εδώ έχουμε μερικά σημαντικά θέματα. Πρέπει να φροντίσουμε να συμφωνήσει και η Επιτροπή Βιομηχανία, να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, αν θέλετε. Πιστεύω ότι οι τροπολογίε μα τουλάχιστον καλύπτουν τα δικά μα θέματα και αυτό προσθέτει αξία και είναι και υπέρ τη ε, Επιτροπή Βιομηχανία. Λοιπόν, ποιο άλλο από τη Γενική Διεύθυνση Enterprise, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο, πείτε μας ε, ποιος είστε και σας ακούμε. Σημαντική καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για το έργο της και την συμβολή της. Περιμένουμε σχόλια και τροπολογίες που ήδη βρίσκουμε σύμφωνα και με τις δικές μας ε, απόψεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριε Κουφεράτη, λοιπόν, έχετε τον, λόγο για να κλείσουμε. Υπενθυμίστε μας αν θέλετε και το χρονοδιάγραμμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό που σας είπα και πριν. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε στις 5 Σεπτεμβρίου. Συνεπώς, ζήτησα και γι' αυτό το λόγο ζήτησα επίμονα από τους συναδέλφους να διαβάσουν το ταχύτερο το σημείωμα που σας έστειλα χτες με τις προτάσεις συμβιβασμού και να μου ζήτησα από τους συναδέλφους να αποστείλουν τις παρατηρήσεις και ενδεχόμενες προτάσεις διόρθωσης το αργότερο μέχρι πέμπτη το βράδυ, διότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος για περαιτέρω συζητήσει. Ε, θα περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία μέσω μιας εργασίας συντακτικής φύσης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό βέβαια για τους λόγους που σας προείπα. Τα οι τροπολογίες που μου αποστήλατε, κατά την άποψή μου, είναι τροπολογίες που είναι συμβατές με το κείμενο, άρα ένα μέρος θα ενταχθεί στις προτάσεις συμβιβασμών και οι άλλες θα γίνουν αποδεκτές ως τροπολογίες καθαρά, διότι σχετίζονται με το γενικότερο θέμα προβολής των θέσεών μας. Άρα κάθε τροπολογία κρίνεται και αν τη συμμεριζόμαστε τότε μπορούμε να την προωθήσουμε ως έχει. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση με βάση τις γνώσεις που έχουμε Και όταν διαβάσετε τις προτάσεις συμβιβασμού θα δείτε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε θετικά σε μια θετική έκβαση στις 5 Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου χωρίς δυσκολίες. Στην, ε, κατά την κατανομή των τροπολογιών, είχαμε την ε, αγαστή συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων δεν ε, προβάλλονται εναλλακτικές. Αυτό δεν ε, συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Συνέβη όμως και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Good. Well, thank you very much uh, indeed. And you gave us... Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μια καλή βάση ώστε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, περιμένουμε 5 Σεπτεμβρίου την ψηφοφορία μέρους και των σχεδόν υπόσχομαι ότι θα στείλουμε εγκαίρως τροπολογίες και συμβαστικές. Λοιπόν, προχωρούμε με το τελευταίο σημείο για σήμερα. Έχουμε χρόνο μέχρι 5 και 4. Ασφάλεια προϊόντων. Έχουμε εδώ τους δύο συζήτητες. Σαλντεμόζε και πείτε Κάινεν. Θεωρώ τις δύο εκθέσεις συναφής. Είναι η κυρία Σπανού εδώ από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ και ο κύριος από την Γενική Διεύθυνση για τις επιχειρήσεις. Ή όχι, ή κάνω λάθος. Έχουμε ασφάλεια λοιπόν καταναλωτικών προϊόντων και υποπτία τη αγορά προϊόντων. Και επιτόντο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και επιτόντο είναι εδώ. Τζιουζιπίδα επιτόντο λοιπόν, τώρα σα είδα. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική ομάδα η οποία θα απαντήσει και θα σχολιάσει τα κείμενα. Έχουμε λοιπόν σχέδια εκθέσεων από δύο ισχύτες. Θα δώσω τον λόγο στις δύο εισηγήτριες, μετά θα συζητήσουμε. Να δούμε ποιοι είναι εδώ από τους Σκιώδης. Μπαλτεσάρη, σκιώδης για την έκθεση Και ο κύριος Κρότσμαν, μετά τον κύριο Φυσιόνι. Είναι ο πλέον σκληρά εργαζόμενος εδώ σήμερα και η κυρία Ρούτερς ε, μεταξύ των γυναικών η πλέον σκληρά εργαζόμενη ο σκιώδης. Και Φόξ, κ. Φόξ μόλι μπήκε στην αίθουσα. Οπότε είμαστε όλοι εδώ, δεν λείπει κανένα από του σκιώδει εξαιρετικά. Ποιο θέλει τον λόγο, ε, σύμφωνα με τον καταλόγο μου, κ. Σαλντεμόζ έχει πρώτη τον λόγο. Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω τις βασικές γραμμές της εκθέσης μου. Να ευχαριστήσω όμως καταρχήν τους Κιώδης με τους οποίους είχαμε διάφορες συζητήσεις εξαιρετικές συζητήσεις και ήδη έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε καλές συμβαστικές τροπολογίες. Δεν έχω αντίρρηση να συζητήσω και κάποιες διατυπώσεις για να διευκολύνω και τους σκιώδεις. Όλα αυτά πολύ καλά. Δεύτερον, είχα την εντύπωση και νομίζω θα συμφωνήσουν από αυτού και οι σκιώδες ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δουλέψουμε στο. το όσο πιο γρήγορα γίνεται για να κλείσουμε το θέμα πριν το τέλος της εντολής. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνουμε υποχωρήσει ως προς την ποιότητα. Συμφωνούμε όμως ότι από εδώ και πέρα θα δουλέψουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Χθε μάλιστα ε, τον Υπουργό Εκπρόσωπο της Προεδρίας είπαμε ότι και αυτοί έχουν διάθεση να εργαστούν σκληρά. Πριν έρθω στα τη. έκθεσης, παρακαλώ Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν για το συγκεκριμένο θέμα, την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, έχει υιοθετήσει πολλές από τις ιδέες μας που είχαμε συμπεριλάβει στην πρώτη μας έκθεση πριν από δύο χρόνια. Υπάρχει δηλαδή ήδη μια καλή κοινή βάση για συζήτηση. Όσο εδώ καλά. Τέσσερα θέματα ουσιαστικά θίγω στην εκθέσή μου, οριζοντίου ενδιαφέροντος. Πρώτον, θεωρώ ότι δημιουργούμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τα καταναλωτικά προϊόντα. όπως έχουμε ήδη κάνει και σε άλλους τομείς. Δεύτερον, όπως ε, είχα πει και σε προηγούμενες συσκέψεις μας, πρέπει να επανεισαγάγουμε την αρχή της πρόληψης. Αυτό το τονίζω σε διάφορα σημεία της έκθεσης. Ίσως έχω επαναληφθεί περισσότερο από ό,τι πρέπει. Θα το δούμε αυτό, θα το λύσουμε. Όμως, είναι μια αρχή που έχει τεράστια σημασία. Οι κατασκευαστές επίσης πρέπει να γνωρίζουν και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού ότι δουλεύουμε με βάση την αρχή της πρόληψης. Αυτό το λέμε βεβαίω σαφώς. Γιατί θεωρούμε την αρχή αυτή ως βασική αρχή. Πίστευε επίση προσωπικώς ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και την αποφασία 768 του 2008. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους ορισμούς στον κανονισμό. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη, παραλαμβάνω, ευθυγράμμιση. Ιδιαίτερα στους ε, τομείς που αφορούν τις υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Τονίζω επίσης την ασφάλεια από το στάδιο του σχεδιασμού. Ασφάλεια κατασκευής. Πάλι σημασία όταν παράγουν προϊόντα η βιομηχανία να λαμβάνουν την ασφάλεια υπόψη τους από την αρχή, από το στάδιο του σχεδιασμού. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που θίγω στην εκθεσή μου. Τώρα σου πω στα ειδικά. Θεωρώ ότι αξίζει να αναφέρουμε και να τονίσουμε την θέση στην οποία βρίσκονται οι καταναλωτές. Την ευπαθή θέση, ιδιαίτερα των παιδιών. Εξαιτία προϊόντων τα οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά. Δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική διατύπωση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ορίσουμε κάπως αυτά τα προϊόντα τα οποία ασκούν ιδιαίτερη έλξη στα παιδιά, να το δούμε και με τους σκιώδεις, αλλά θέλω αυτό το μήνυμα να φτάσει στην βιομηχανία, όχι μόνο στις αρχές. θεωρούν ότι το έχουμε ρυθμίσει το θέμα. Αλλά πιστεύω ότι το θέμα πρέπει, το μήνυμα μάλλον να φτάσει και στην βιομηχανία, στους κατασκευαστές τέτοιου είδους προϊόντων. Τι είναι αυτά λοιπόν τα ιδιαίτερως ελκυστικά προϊόντα για τα παιδιά. Ε, χρειαζόμαστε, όπως είπα, έναν ορισμό. Επίσης, μπορούμε να και πρέπει να θεσπίσουμε ένα πιο προηγμένο σήμα, CE, ένα κοινωτικό σήμα, CE+, CE, συν. Ένα πράγμα το οποίο παραπλανά συνήθω του καταναλωτέ είναι η ύπαρξη του σήματο που κάνει πολλού να πιστεύουν ότι πρόκειται για δοκιμασμένο προϊόν. Αυτό δεν ισχύει. Οπότε είτε θα πρέπει να αποσύρουμε πλέον το σήμα ή e από τα προϊόντα ή θα εισαγαγούμε ένα νέο σήμα, C+, με το πρόσημο συν δηλαδή, το οποίο αυτό ακριβώς θα σημαίνει ότι το προϊόν είναι δοκιμασμένο από κάποιες αρχές. Αυτό θέλει προσεκτική συζήτηση. Και εδώ νομίζω ότι εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές με την κίνησή μας. Να το συζητήσουμε παρακαλώ αυτό. Όχι αναγκαστικά σήμερα, αλλά το λέω γιατί κάποιε αρχέ επιτήρηση τη αγορά πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά από την πλευρά των καταναλωτών εδώ έχουμε, οφείλουμε να κάνουμε κάτι. Επίση, να δούμε το θέμα των κυρώσεων. Πρέπει να γίνουν αυστηρότερε, να οργανωθούν και να έχουν αποτέλεσμα. Να είναι δηλαδή αποτρεπτικέ όσον αφορά τι απάτε που κάνει η βιομηχανία. Να παράγει τέλει ασφαλή προϊόντα. Πιστεύω επίσης ότι είναι από τα πιο επίμαχα ζητήματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα αφορά την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την ένδειξη της προέλευσης. Νομίζω ότι θα είναι το παρελθόν ένα καυτό θέμα. Στην έκθεσή μου δηλώνω ότι πιστεύω ότι είναι καλή η ιδέα να αναφέρεται η προέλευση. Υπάρχει ένδειξη της προέλευσης το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει, κατά παράληψη μάλιστα, ένα βελτιωμένο σχήμα. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους καταναλωτές, όχι μόνο για τους σκοπούς της χρηλασιμότητας, γιατί κατά τα υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που επιτρέπουν την, τον προσδιορισμό της προέλευσης. Όμως, χάρη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει η βιομηχανία, οι κατασκευαστές να βάζουν μια διεύθυνση πάνω στο προϊόν, που πολλέ φορές όμως μπορεί να είναι παραπλανητική έτσι όπω. έχουν τα πράγματα σήμερα. Ας πάρουμε μια ταινία, μια επιχείρηση από τη Δανία, η οποία έχει την έδρα της στη Δανία. Η διεύθυνση που θα εμφανίζεται θα είναι στην Κίνα, αλλά το προϊόν μπορεί να προέρχεται από την Κίνα ή κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καταναλωτή ο οποίο διαβάζει μια διεύθυνση στη Δανία, μπορεί να παραπλανηθεί και να πιστέψει ότι το προϊόν είναι από τη Δανία. Αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Η ένδειξη λοιπόν προέλευση πρέπει να είναι χρήσιμη, να μην παραπλανά. Αυτό θέλω να συζητήσουμε παρακαλώ. Όπως είπα και στου ε, εισηγητέ, το λέω και σε εσά τώρα, ίσως να πρέπει να βρούμε μια λύση με την οποία θα ευθυγραμμίζεται η απέτηση στην Ευρώπη με αυτές στις ΗΠΑ όσον αφορά την ένδειξη προέλευσης. Υπάρχουν πολλές εταιρείε που παράγουν ούτως ή άλλως για τις ΗΠΑ, άρα η απέτηση αυτή δεν ε, αποτελεί πλέον επιβάρηση. Αν πάρετε ένα iPhone θα δείτε ένα iPhone είναι συναρμολογημένο στην Καλιφόρνια αλλά παράγεται στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τι επιχειρήσει, αλλά θέλουμε να έχουμε μια σαφή ιδέα της προέλευσης. Το λέω αυτό, διότι ήρθε ο καιρό να στείλουμε το μήνυμα ότι θέλουμε να ξέρουμε πού φτιάχνουν τα προϊόντα. Να γίνουμε με τρόπο ο οποίο δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τις επιχειρήσεις. Τρίτον, και τέλο για το θέμα αυτό, πιστεύω ότι έχει σημασία να μην ξεχνούμε ότι 10% των σημάτων των ειδοποιήσεων αφορά προϊόντα των οποίων δεν είναι γνωστή προέλευση. Σε αυτή την περίπτωση οι αρχέ δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει. Τέλο, γενικότερα, θέλω να πω ότι εγώ προσωπικώς θα ήθελα να κάνω μια προσπάθεια να βρούμε έναν τρόπο να θυρανίσουμε, να εναρμονίσουμε, αν θέλετε, τις προσπαθίες μας στο διατλαντικό επίπεδο. Να εναρμονίσουμε τις προσπαθίες μας εμείς και οι ΗΠΑ. Κάπου είναι καλύτεροι οι Αμερικανοί, κάπου εμείς. Αυτόν τον κύριο βεβαίω είναι πολύ τη μόδα και οι συζητήσει για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τι ΗΠΑ. Θα ήταν λοιπόν ακόμη περισσότερο χρήσιμο να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε και το δικό μας νομοθέτημα, να λάβει υπόψη το ακριβώ την επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι να συμβαστούμε, όχι να κάνουμε βήματα πίσω εις βάρος των καταναλωτών, αλλά το αντίθετο. Με αυτά, ξαναλέω ότι προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία, ανάψη του νέου νομοθετήματος, Έχω διάθεση να τροποποιήσω αν χρειαστεί διάφορες διατυπώσεις βάσει και των τροπολογιών. Πάντως το πιο σημαντικό είναι να δηλώσουμε ότι το θέμα είναι σημαντικό. στόχος μας είναι περισσότερη ασφάλεια για τους καταναλωτές και ισότιμη κανόνε βεβαίω για όλου του κατασκευαστέ. Ισορροπία μεταξύ και των δύο. Αυτού του δύο στόχου θέλουμε να συγκεράσουμε και γι' αυτό και θα δεχθώ τροπολογίε. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι χρήσιμο για όλου και το οποίο θα οδηγήσει και σε μια πιο λειτουργική εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, πολύ εκτεταμένη άποψη και παρουσίαση που μας κάνετε και για το πού θέλετε να γίνουν οι αλλαγές. Πολύ καλό αυτό. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πιετικάνιεν, γιατί νομίζω ότι θα ακούσουμε τα δύο θέματα αυτά και θα συζητήσουμε από κοινού. Και μετά, κυρία Σαλντεμόζα, είσαστε σκιώδες για το θέμα της κυρίας Πιετικάνιεν, οπότε αν θέλετε πάλι το λόγο θα σας το ξαναδώσω. Κυρία Πιετικάνιεν. Ευχαριστώ πάρα πολλά και, πολύ και νομίζω ότι όντω να είναι πολύ λογικό να συζητηθούν από κοινού τα δύο θέματα αυτά είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, ε, ο κανονισμός και μετά η εφαρμογή. Καταρχάς, να πω ότι πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ καλή, είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Βελτιώνει σημαντικά την κατάσταση όπως έχει σήμερα. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πολύ κατακριματισμένη η αγορά και ότι τα εθνικά συστήματα Και ξέρουμε επίση ότι μόνο 0,3% όλων των προϊόντων που εισάγονται διατίθενται στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχονται από τι αρχέ. Χρειάζεται λοιπόν α, καλή συνεργασία και η πρόταση είναι καλή γενικά ω αρχή. Και παρά το γεγονό ότι άλλαξε από οδηγίε σε κανονισμό, μας ε, προκαλεί κάποια επιπλέον ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν με το Συμβούλιο για θέματα εποπτείας. Ο ορισμός του κινδύνου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε τον κίνδυνο με πιο ευρύ τρόπο προκειμένου να διευκρινίζει και θέματα ασφάλειας αλλά και μη συμμόρφωσης. Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και οι κανονισμοί που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για τη συμμόρφωση των αγορών που εισάγονται στην αγορά μας. Άρα τα προϊόντα τα οποία είναι επιζήμια, επιβλαβή, αλλά και τα προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονται με διάφορες διατάξεις ασφαλείας και λοιπές διατάξεις. Φυσικά αυτό είναι σημαντικό από πλευράς κινδύνου αφενός, είναι όμως και σημαντικό και από πλευρά του καταναλωτή και σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των παραγωγών και τους ε, ίσους όρους λειτουργίας. Ως τώρα δεν έχω ακόμα ακούσει αρνητικά σχόλια για το θέμα αυτό, αλλά θα ήταν σημαντικό. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σχολιάσει. Ένα άλλο σημείο το οποίο αποτελεί μεγαλύτερη αλλαγή επί της ουσίας είναι οι διοικητικέ κυρώσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα αποθάρρυνση σε ό,τι αφορά τη μη συμμόρφωση. Τι προτείνεται διοικητικές κυρώσεις έως και 10% του κύκλου εργασιών αλλά σε περίπτωση σοβαρής ε, δόλειας παραβίασης των κανονισμών. Έλαβα σχόλια ότι ενδεχομένως να είναι πιο σωστή η σύνδεση με το κέρδος που προκύπτει από την πώληση του προϊόντος και όχι τόσο με τον κύκλο εργασιών του, της επιχείρησης γιατί μπορεί να είναι μια εταιρεία η οποία να παράγει πολλά προϊόντα. Να ακούσω τα δικά σας σχόλια για το θέμα αυτό. Ένα άλλο θέμα το οποίο ακόμα δεν έχω προτείνει, το έχω αφήσει ανοιχτό, ε, ζήτησα από τους κοιότες να το σχολιάσουν, είναι πώς μπορούμε να ε, επιτρέψουμε να συμμετέχουν και τα κέντρα των καταναλωτών. Αυτό όχι για να μειώσει την επίσημη ευθύνη των αρχών, αλλά αν συμμετέχουν καλύτερα οι ενώσεις και τα κέντρα καταναλωτών, οι καταναλωτές θα είναι πιο σωστά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους, για το τι σημαίνει η ασφάλεια προϊόντος ή για το ποιες είναι οι δυνατότητες επικοινωνίας με τους αρμόδιους δημόσιους υπάλληλους. Ενδεχομένω να υπάρξουν κάποιε σχετικέ εκστρατείε και θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε σχετικά με το θέμα αυτό. Τέταρτο σημείο. Το φόρουμ για την, ε, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Εποπτεία Αγορά. Για την ενέσχυση του ρόλου τη και τον συντονιστικό του ρόλο. για αρχές που ενδεχομένω να μην ε, εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Τελευταίο στοιχείο, και δεν προτείνω να τροποποιηθεί εδώ σε αυτόν τον κανονισμό, αλλά σε άλλη διάταξη, να αναπτυχθεί μια νέα μέθοδος για να βελτιωθεί η εποπτεία της αγοράς. Γιατί ιδιαίτερα στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η διεύρυνση του δεμπορίου που είναι φατικό στοιχείο, Δεν βλέπω να μπορούμε να ε, κάνουμε εντελεχείς ελέγχους από δημόσιους υπαλλήλους. Και θα ήταν τόσο κοστοβόρο για τους παραγωγούς να κάνουν τέτοια, τέτοιους ελέγχους στα σημεία ελέγχου, στα σημεία εισόδου. Αν, για παράδειγμα, αυξάναμε το ποσοστό ελέγχου σε 30%, που ούτε αυτό θα ήταν σωστό. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικές λύσεις και να τις εξετάσουμε σοβαρά προκειμένου να μην αυξηθεί το διοικητικό άχθος, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και τι προτείνω στο σημείο αυτό. Στην αναθεώρηση να ξεκινήσουμε ένα σύστημα ελέγχου από τρίτα μέρη. Έχουμε κάποια εμπειρία από τέτοια συστήματα ελέγχου, όχι μόνο σε θέματα λογιστικά, σε κάποια κρατημέλη όπου υπάρχουν συστήματα σε καλές εταιρείε πάντα υπάρχουν εσωτερικά συστήματα ελέγχου ποιότητας και αυτές οι, οι καλοί, οι έχουν εξωτερικούς ελεγκτές για να ελέγχουν τα συστήματα ποιότητάς τους, αλλά για να κάνουν τεχνολογικούς ελέγχους για την ποιότητα των προϊόντων. Άρα, αν καθίστανται υποχρεωτική αυτή η έλεγχη, το επιπλέον κόστος θα ήταν μεγάλο, δεν θα είναι μεγάλο, αλλά θα σήμαινε για τις ε, επιχειρήσεις που έχουν ενδεχομένως επικίνδυνα προϊόντα μεγάλη βελτίωση. Και έτσι θα είχαν ίσους όρους όλες οι εταιρείε. Και αυτό που θα κάναμε στη συνέχεια αν ήταν ένα μελλοντικό υποχρεωτικό σύστημα, να υπάρχει εσωτερικός αλλά και εξωτερικός έλεγχος υποχρεωτικά και να μην επιβάλλονται κυρώσεις τόσο στον παραγωγό αλλά στον ελεγκτή. Αυτό γίνεται ήδη σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στον χρηματοοικονομικό κλάδο. ό,τι αφορά για παράδειγμα οίκους αξιολόγησης που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εφαρμόσουμε ένα ανάλογο σύστημα προκειμένου να γίνεται έλεγχος από εταιρείε που έχουν κάποια κατάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα τους προέτρεπε να κάνουν σωστές, σωστούς ελέγχους, θα τους απέτρεπε από λανθασμένες ε, τέτοιους ε, ελέγχους και έχω ακούσει πάρα πολλές φρικτές ιστορίες για χημικά τα οποία ε, λαμβάνουν άδεια κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούνται στην κλωστοφαντουργία και δημιουργούν τελικά, παράγουν προϊόντα που δεν είναι ασφαλή. Αυτό που λέω είναι ότι όταν ένα προϊόν κοστίζει 9 ευρώ και ένα αντίστοιχο κοστίζει 90, μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος για τη διαφορά τιμής αυτή. Αυτά λοιπόν τα σχόλια μου για το θέμα αυτό. Λυπάμαι μακρηγόρησα, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπηρετήσατε πολύ καλά αυτό το σκοπό. Έχουμε μέχρι τις 5 και 4 και χαίρομαι για τον ενθουσιασμό σας. Το θέμα αυτό έχει ένα τίτλο που δεν αντικατοπτρίζει την σημασία του πραγματικά για τους πολίτες. Κυρία Σάλντεμόζε, θέλετε να επανέλθετε στο τέλος. Ωραία. Μπαλντασάρι. ο Σκιώδης. Μετά, Κρόιτσμα. κυρία Ρούλε και ο κύριος Φόξ. Και όποιος άλλος το επιθυμεί, ο κύριος Μπαλντασάρι. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τις ε, δύο εισηγήτριες για το ότι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το πολυσχηδές ε, σχήμα που αφορά την εποπτεία των προϊόντων της αγοράς. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, ιδιαίτερα σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων γιατί είμαι σκιώδης για τη συγκεκριμένη έκθεση. Σημερίζομαι τις γενικές αρχές της εισηγήτριας για απλούστευση και συμπλήρωση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας επί του θέματος και δημιουργία ενός δικτύου, δικτύου ασφαλείας όπως όρισε η εισηγήτρια για να υπάρχει μία οριζόντια αντιμετώπιση του συστήματος ε, εποπτείας και προστασίας των προϊόντων. Θα ήθελα όμως να σταθώ και ένα άλλο ζήτημα. Εάν λάβουμε υπόψη και τα εναρμονισμένα προϊόντα, θέλουμε να πληρώσουμε αυτό το κενό του συστήματος και θα θέλαμε να μην καταστούν ορισμένοι τομείς υπερρυθμισμένοι και άλλοι όχι τόσο. Άρα αυτό το δίχτυ ασφαλείας θα πρέπει να καλύψει τα χάσματα του συστήματος χωρίς να επιβάλλει επιπρόσθετο κόστος στους τομείς που έχουν ήδη ρυθμιστεί. θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπως αναφέρθηκε. Η αρχή της προειδοποίησης θα πρέπει να σχετίζεται και με τον ορισμό που ορίζει το ΔΕΚ. Ίσως υπάρχει μία ε, διακριτική ευκαιρία, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές αποτιμήσεις από, την, ε, από τις αρχές εποπτείας. Δεν θα πρέπει στις διάφορες χώρες να υπάρξει διαφορετική εφαρμογή αυτής της αρχής, δημιουργώντας ε, στρέβλωση της αγοράς και αθέμητο ανταγωνισμό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτή η πτυχή του θέματος. Δέχομαι την επέκταση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ως προς το σήμα συμφωνώ με την προστιθέμενη αξία, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι δεν θα πρέπει να σημαίνει αυτό επιπρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις και δέχομαι και τις ευάλωτες κατηγορίες που προαναφέρθηκαν, αν και στη φάση του προγραμματισμού χρειαζόμαστε ένα καλύτερα προσδιορισμένο κριτήριο. Πολλές φορές αυτή η ευαλωτότητα ορισμένων προϊόντων σχετίζεται, από σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει διαφορετική αποτίμηση. Με αυτή την οδηγία προσπαθούμε να ορίσουμε ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι το θέμα της ευθύνης των κατασκευαστών και των διανομέων και θεωρώ ότι η αρχή της προέλευσης θα πρέπει να ενταχθεί σε μια λογική, στη λογική της μεγαλύτερης ασφάλειας. Δεν μπορούμε να έχουμε υψηλότερη ασφάλεια για τον καταναλωτή αν δεν ε, χορηγούνται πληροφορίες. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι η παροχή πληροφοριών. Όσο περισσότερο γνωρίζει την πορεία του προϊόντος ο, ο καταναλωτής, τόσο είναι σίγουρος για την ασφάλειά του. Ελπίζω λοιπόν ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και πέντε χρόνια πριν, δεν θα πρέπει να ανοίξουμε νέα κεφάλαια, δηλαδή ε, νέους να ε, προβάλλουμε και να δώσουμε νέες μάχες με σκέψεις που δεν έχουν ε, απόδειχτη, γιατί μιλάμε για διοικητικό κόστος κλπ. Όλα αυτά δεν έχουν απόδειχτη. Γι' αυτό το θέμα της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί στην περίπτωση του, των ΙΠΑ, του Καναδά, ε, της ε, Κίνας και της Ιαπωνίας δεν μπορούμε να αναφέρθουμε σε τίποτα Δηλαδή, αγοράζουν ε, παρμιτζάνο δίθεν προέλευση, το οποίο δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση με το παρμιτζάνο ρετζάνο. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το τομέα. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και χωρίς ε, ιδεολογικές μάχες. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει να δούμε και το turnover και το κύκλο εργασιών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και τα προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο ε, σίγουρα. Ασφαλή δηλαδή. Ωραία, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος για την άποψή σας και για το ε, ε, πάθος σας σε σχέση με την προέλευση ορισμένων προϊόντων. Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις δύο εισηγητρίες. Θα αναφέρω και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Από κοινού. Το σήμα C+. Η πρόταση να αντικατασταθεί το μέση Plus βάσει ελέγχου τρίτων ανεξαρτήτων ομάδων μας θυμίζει την πρόταση του συναδελφού ΣΒΑΠ του 2007. Μια τέτοια πρόταση της κυρίας Σαλδεμόσα θα μας έβρισκε σύμφωνους. Αλλά μόνο εάν είναι σε εθελούσια βάση και υπόκειται σε υψηλές προδιαγραφές, εξίσου υψηλές με αυτές των εθνικών ε, προδιαγραφών. γιατί δεν έχει νόημα να είναι κάτω από το επίπεδο των ε, εθνικών αγορών. Δυστυχώς πριν από έξι χρόνια δεν καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία για ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σήμα. Είμαι σκεπτικιστικός δηλαδή, αλλά δεν είμαι επί της ε, αρχής ε, αντίθετος. Η εισαγωγή εθνικών σημείων επαφής είναι ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί και στην πράξη. Ειδικότερα αναρωτιόμαστε, θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες οι οποίες θα κοστίζουν Ίσως μέσω των εμπορικών επιμελητηρίων θα μπορούσαμε να κινηθούμε και να σκεφτούμε κατά πόσον χρειαζόμαστε χρηματο, χρηματική χρηματοδότηση. Είναι πολύ στενά τα περιθώρια και δεν έχουμε πολλά χρήματα, πολλά κονδύλια. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ε, κυρώσεις, τις ποινές, για το ποσοστό του κύκλου εργασιών, για το ποσοστό επί των κερδών του συγκεκριμένου προϊόντος. Το θέμα είναι να είναι εξαιρετικά αναλογικές ε, οι κυρώσεις. Είτε πρόκειται για τον κύκλο εργασιών του συνολικό, είτε για τον κύκλο εργασιών του συγκεκριμένου προϊόντος. Γιατί το θέμα δεν είναι να φαλυρίσει η εταιρεία. Μπορούμε να ορίσουμε ε, μια χρηματική ποινή επί του συνόλου του κύκλου εργασιών, να το σκεφτούμε βάση περιπτώσει. Και τώρα να περάσω στα αρνητικά και να περάσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφο Μπαλτασάρη. Κύριε Μπαλτασάρη, είναι δυνατό να πιστεύετε και εσεί ο ίδιο ότι το προϊόν όταν είναι made in China, όταν αναφέρεται έχει να κάνει με την ασφάλεια του προϊόντος, είπε και η κυρία Σαντεμόζα, είναι σχεδιασμένο στη ΣΥΠΑ, αλλά κατασκευασμένο στις, στην Κίνα. Μα δεν λέει τίποτα το γεγονός ε, στον καταναλωτή του τι αναφέρεται που είναι κατασκευασμένο το προϊόν. Να πιστεύουμε ότι για την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων ότι η, η αναφορά της χώρας που κατασκευής ε, είναι εγγύηση ποιότητας, αυτό τι να πω είναι χήμερα. έχω και ένα ωραίο παράδειγμα να σας αναφέρω. Όχι αυτό που είπε η κυρία Σαλτεμόζο, νομίζω ότι είτε η Samsung είτε κάποιος άλλος, ε, κάποια άλλη κατασκευάστρια που παράγει στην Τσεχία αναφέρει ότι παράγεται στην Τσεχοσλοβακία και θα έπρεπε να λέει κατασκευάζεται στην Τσεχοσλοβακία αλλά αν είναι παραπάνω το ποσοστό από 40% ε, παράγεται στην Κίνα, θα πρέπει να φέρετε παράγεται στην Κίνα. Όταν μιλάμε για διεθνώς ε, κατασκευασμένα προϊόντα, φυσικά μας ενδιαφέρει ένα γνωστό όνομα να είναι ασφαλές, ανεξάρτητα από το αν κατασκευάζεται στην Κίνα, στη Φιλανδία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. γιατί θα ήταν μεγάλο πλήγμα και για την εικόνα ακόμα της εταιρεία αν δεν ήταν ασφαλές το προϊόν. Και λέει ο κ. Μπαλτασάρε ότι φυσικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει αυτό το σύστημα εντοπισμού και αυτό συνεπάγεται μεγάλη γραφειοκρατία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αυτό που είπε η κυρία είναι σωστό. Θα πρέπει να μην δυσκολεύουμε τις επιχειρήσεις μας εδώ στην ε, Ευρώπη, προκειμένου να φεύγουν ακόμα πιο πολλές εταιρείε με τέτοια θέματα ανιχνευσιμότητας και με τέτοια θέματα σήμανσης. Θα πρέπει όλα να τα ρυθμίσουμε. Τώρα, αυτό θα πρέπει να ισχύει για τα εναρμονισμένα προϊόντα και δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξουμε και κάποια προϊόντα που εξαιρούνται. Έχουμε τα συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο κανονισμό και το γενικό κανονισμό. Αυτό δημιουργεί γενικώ μια, μια σύγχυση και θα έπρεπε να τα αποφύγουμε αυτό. Τώρα για την έκθεση ποιοτικά είναι. Σε γενικέ γραμμέ είναι καλή, θα επικεντρωθώ μόνο στα αρνητικά, ε, κυρία συνάδελφε. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα θετικά. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην θεωρούνται αυτόματα επικίνδυνα όλα τα προϊόντα που δεν είναι απόλυτα συμβατά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και αυτό δεν αναφέρθηκε ε, επαρκώς. Δεν θέλουμε φυσικά επικίνδυνα προϊόντα, αλλά τι είναι το προϊόν που δεν είναι συμβατό, που δεν συμμορφώνεται. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια ε, διαφοροποίηση, γιατί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναφέρονται ως RAPEX όλα τέτοια προϊόντα που ενδεχομένως να είναι επικίνδυνα, θα σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την κατηγορία και προϊόντα τα οποία ενδεχομένως έχουν μια μικρή μη συμμορφώση. Και ίσως αυτά τα προϊόντα θα έπρεπε να αναφέρονται στη βάση δεδομένων ESM για να μην υπερβα... Ε, υπε... επιβαρυνθεί υπερβολικά το RAPEX και θεωρούνται όλα αυτά τα προϊόντα επικίνδυνα. κοιτώντας ότι για παράδειγμα ένας παραγωγός πρέπει να κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και το τι σημαίνει αυτό για τον έλεγχο, νομίζω ότι γενικά θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή της αναλογικότητας ό,τι αφορά και αυτό το θέμα. Η μερική ή συνολική χρηματοδότηση της εποπτείας της ε, αγοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρηματολογείται από τη φορολογία. Εάν είναι να αρχίσουμε να κάνουμε διακρίσεις, καλύτερα να το καταργήσουμε το σύστημα. Και δεν ξέρω αν κάτι αυτό συνταγματικό στη Γερμανία. δεν υπάρχει και σωστή ανάλυση των κινδύνων. Και εδώ θα ήθελα λοιπόν αυτή η παράγραφος να διαγραφεί και τώρα να περάσουμε στις χρηματικές ποινές. Τουλάχιστον 10% του κύκλου εργασιών. Το θέμα είναι γιατί τι μέγεθος μιλάμε. Ας υποθέσουμε ότι έχει κανείς, για παράδειγμα, μισό ή 1% κέρδος. Αν είναι υπερβολικό, υπερβολική η ποινή, το καθοριστικό είναι ο παραγωγός. Δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε την ευθύνη από τον παραγωγό. Ιδάλλως όλο το επιχειρηματικό μοντέλο θα καταρρεύσει. Αυτά λοιπόν γι' αυτό επικεντρώθηκα στα πιο αρνητικά και τα καλά τα θετικά δεν τα ανέφερα και στις δύο εκθέσεις. Ασφαλώς υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια θετικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Πολύ επικοδομητικά τα σχόλια. Να μην επαναλάβουμε βεβαίω πρώτα ε, που έχουμε πει. Νομίζω ότι θα βρούμε. Η κυρία Ρούλα να ευχαριστήσω τις ηγητρίες για την καλή συνεργασία, γιατί νομίζω ότι πραγματικά θα βρούμε μια καλή λύση, την οποία θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλοι. Ωστόσο θα ήθελα... Ωστόσο θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερως. Θα πρέπει να κοιτάξουμε του ορισμού. Δεν είναι νομίζω σωστό υπό τον όρο κίνδυνο να περιλαμβάνονται και θέματα συμμόρφωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση αφενό μεταξύ τη συμμόρφωση και αφετέρου μεταξύ του κινδύνου. Να εξηγήσω να δώσω το παράδειγμα της κυρίας Σάλντεμόζα με το σήμα CE, το οποίο τι σημαίνει ότι είναι κανείς συμμορφωμένος και συμφωνώ ότι δεν το χρειαζόμαστε αυτό γιατί πάντα το ερμηνεύει ε, λάθος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανείς δεν το σκόπευε φυσικά αυτό, δεν είχε αυτό σκοπό. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως θα πρέπει να το καταργήσουμε τελείως αυτό το σήμα. Σε καμία περίπτωση όμως όταν δημιουργήσουμε, αν δημιουργήσουμε ένα δεύτερο σήμα και θεωρήσουμε τον παραγωγό υπεύθυνο για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων να το ονομάσουμε C+, γιατί αυτό θα ενίσχυε περαιτέρω αυτή την ε, παρεξήγηση. Θα έπρεπε να βρούμε ένα νέο σήμα, θα πρέπει να σκεφτούμε ασφαλώς πώς θα πρέπει να αυξήσουμε την ευθύνη του παραγωγού για προϊόντα τα οποία απευθύνονται σε ευάλωτους καταναλωτές. με μεγάλο βαθμό επικίνδυνοτητάς υπάρχει το σύστημα τρίτης ε, πιστοποίησης, πιστοποίησης τρίτου να υπάρχει για παράδειγμα και μια διαχείριση ποιότητας μέχρι να γίνει τέτοιο έλεγχος. Πολλές φορές το κάνει αυτό μια εταιρεία χωρίς να υπάρχει επιπλέον κόστος. Να το σκεφτούμε και αυτό. Αλλά αυτά θα λειτουργήσουν μόνο αν υπάρξει διάκριση μεταξύ συμμόρφωσης και ασφάλειας. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Να μην υπάρχει πάλι τέτοια σύγχυση. Τώρα, θεωρώ ότι υπάρχει μια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα περάσει αυτό από το Συμβούλιο, αλλά να πω το εξή. Η αρχή της χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να υπερεπιβληθεί σε ό,τι αφορά θέματα ασφάλειας και να μην επιβαρυνθεί επίσης υπερβολικά και να την προσπαθήσουμε να το χρησιμοποιήσουμε, να τη χρησιμοποιήσουμε για την ανιχνευσιμότητα. Όχι, μιλάμε για ένα θέμα προστασίας ε, θέσεων εργασίας. Ξέρω ότι είναι άλλο αυτό το θέμα και είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, αλλά αυτό προστατεύει τις θέσεις εργασία σε πρώτη φάση και τίποτε άλλο. Η αρχή της χώρας προέλευσης, το country of origin. Να κοιτάξουμε και τι ενδεχομένως να περάσει από το Συμβούλιο γιατί θα ήταν κρίμα να μπλοκαριστεί ο κανονισμός μόνο και μόνο για αυτό το λόγο στο Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποιο τρόπο να αποφύγουμε τους ιδεολογικούς πολέμους, κύριε Βαλτασάρη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Πιστεύω ότι σωστό είναι να καλυφθούν, να πληρωθούν τα κενά. Και σωστό θα είναι να μην υπάρχουν ε, σχετικέ εξαιρέσει. Αλλά συμφωνώ και με τον κύριο Μπαλτασάρη θα πρέπει να προσέξουμε γιατί σε κάποιους ε, τομεί δεν θα πρέπει να καταλήξουμε σε υπερρύθμιση. Να σα ε, πω στο θέμα της αρχής προφύλαξης. Σας υποστηρίζω απόλυτα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αναφερθεί και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή άλλες οδηγίες περιορίζονται στο πεδίο εφαρμογή τους, σωστό είναι να φροντίσουμε να υπάρχει σαφήνεια και να ξέρει ο παραγωγός τι πλήττεται. Θα πρέπει να γίνει διάκριση, όπως σας είπα, μεταξύ επικίνδυνων προϊόντων Έχουμε για παράδειγμα ε, διάφορα τέτοια παραδείγματα σε ό,τι αφορά τρόφιμα, σε ό,τι αφορά παιχνίδια για τα παιδιά. Όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν υπόψη. Υπάρχουν πηγές κινδύνου. Συμφωνώ. Για τις κυρώσει ε, πολλοί μίλησαν για θέματα και για το τελευταίο στοιχείο, το οποίο το έθιξε και ο κ. Κρόιτσμαν, το θέμα της εποπτείας της αγοράς. σε ό,τι αφορά ασφάλεια και συμμόρφωση. Και πάλι υπάρχουν δύο συστήματα. Καταρχάς το σύστημα RAPEX, το οποίο συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ρόιτσμαν, είναι για επικίνδυνα προϊόντα και όχι για άλλα προϊόντα. Ιδάλλως έχουμε και το σύστημα ICSMS σύστημα πληροφόρηση και για την επιτροπή τη αγορά. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει αυτό και πραγματικά εγώ θα υποβάλω σχετικέ τροπολογίε για να τα επανεισάγω αυτά τα στοιχεία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ του κινδύνου και τη συμμόρφωση. Μόνο τότε θα έχουμε μια σαφή γραμμή σε αυτή την έκθεση. Thank you very much. Mr. Fox. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Fox. Πρόεδρε, αρχίζει να γίνεται πολύ παραγωγική ημέρα. Τροπήσαμε ήδη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί πολίσεων. Ε, θα δουλέψω με τους σοσιαλιστές με πολύ χαρά επί του θέματος. Πάντως για τα ασφάλεια των προϊόντων. Ευχαριστώ την κυρία σα για την εξαιρετικά συνεργατική της προσέγγιση. Εγώ να πω δύο λόγια για τα θέματα που πραγματικά εκκρεμούν γιατί για τα άλλα συμφωνούμε όσον αφορά την επέκταση του αντικειμένου του πεδιοφαρμαγής. Εδώ λέει τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσία είναι ασαφέ και πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Έχουμε ζητήσει από την νομική υπηρεσία, θυμάστε, μια διευκρίνηση. Τι καλύπτει αυτό, τι περιλαμβάνεται εδώ και συμφωνώ. Δεν θέλουμε εδώ να δημιουργήσουμε προβλήματα στι επιχειρήσεις. Όσον αφορά την ένδειξη προέλευσης, ένα από τα επίμαχα ζητήματα. Εγώ δεν έχω καταλήξει, η ομάδα μου, η ECR, ούτε αυτή έχει καταλήξει. Θα λέγαμε στο το εξή. Εάν θέλουμε, εάν τελικώ υποστηρίξουμε τη λύση αυτή, πρέπει να είναι υπέρ ασφάλεια, ένα μέτρο υπέρ τη και όχι ένα μέτρο προστατευτισμού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο τελικώς θα βαίνει υπέρ της ασφάλειας των καταναλωτών. Όπως είπα πάντως δεν έχουμε ακόμη σχεδιά συγγνώμη. Όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία προσωμιάζουν με τρόφιμα. Και εδώ, ε, ας πούμε, ε, τι γίνεται με ένα σαπούνι το οποίο έχει σχήμα κέικ, πρέπει να απογορευτεί. Εδώ κίνδυνος είναι μεγάλος. Βεβαίως τη στιγμή που θα το δοκιμάσουν μια φορά, θα ξέρουν ότι αυτό δεν είναι κέικ. Ε, λοιπόν, ό,τι να κάνουμε εδώ, να το κάνουμε βάση του πραγματικού κινδύνου. Γιατί τα παιδιά, αν το δοκιμάσουν, είναι βέβαιο ότι θα το ξαναδοκιμάσουν. Επίσης, για τα ιδιαίτερως ελκυστικά προϊόντα για τα παιδιά. Κατανοώ ότι επιδιώκει η εισηγητρία, όμως φοβούμε ότι εδώ κινδυνεύουμε να θερτήσουμε και εν τέλει ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να απαγορεύσουμε και χωρίς να βελτιώσουμε τις συνθήκες ασφάλειας. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να περιγράψουμε καλύτερα τα επικίνδυνα αυτά προϊόντα. Τώρα για το σήμα, την ένδειξη CE με το πρόσημο SIN δεν συμφωνώ γιατί δεν νομίζω ότι προσθέτει τίποτα ούτε θίγει τον πυρήνα του προβλήματος που είναι η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσει ασφάλεια. Ακόμη και σήμερα, οποιοδήποτε θέλει, βάζει ένα σήμα C ή e πάνω σαν προϊόν και παραπλανεί τον κόσμο. Το ίδιο μπορεί να κάνει αύριο το πρωί κάλλιστα με το CE+. Το θέμα είναι λοιπόν οι μηχανισμοί επιτήρησης της αγοράς για να δούμε τι θα γίνει με τα επικίνδυνα προϊόντα. Επίσης, αρχή της πρόληψης, η προληπτική προσέγγιση. Ήδη αυτό περιλαμβάνεται στις συνθήκες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παραλάβουμε τίποτα εδώ. Η δική μας έμφαση πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση κινδύνου και στις τεχνικές προσεγγίσεις. Κύριε Κρότσμαν, όταν τελειώσετε πείτε μου να συνεχίσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τεχνική φάκελη. Απογοητεύτηκα γιατί δεν λέμε τίποτα στην έκθεση για τους τεχνικούς φακέλους. Πιστεύω ότι η δεκατής περίοδος δεν μας καλύπτει. Στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, σίγουρα πάνω αυτοκίνητα, τα οποία τα κρατάει περισσότερο από 10 χρόνια, αλλά για ένα στυλό και για τις απαιτήσει για τους εισαγωγείς. Δεν νομίζω ότι εδώ πάμε πουθενά. Δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Πρέπει να τροποποιήσουμε την νομοθεσία με τρόπο αναλογικό χωρίς να περιπλέξουμε τα πράγματα για τις επιχειρήσεις. Και δύο λόγια για την βαπτία της αγοράς. Και το λέω αυτό στην κυρία Τικένεν. Υπάρχουν σημεία στα οποία δεν έχουμε ακόμη συμφωνήσει όντως για την αναφορά στα ευρωπαϊκά όργανα. Είμαι υπέρ τη διαφάνεια, αλλά εδώ ζητάει πολλέ λεπτομέρειε και συγκεκριμένα φοβούμε. Με αποτέλεσμα να κάνουμε τη ζωή δύσκολη στι επιχειρήσει. Είμαστε υπέρ μια ισόρροπη προσέγγιση, αλλιώ δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε στο Συμβούλιο για την βάση δεδομένων RAPEX. Ο σκοπό είναι να καταγράψουμε τα σοβαρού κινδύνου. Ναι λοιπόν στην αποτελεσματικότητα, ναι στην καταγραφή των πιο επικίνδυνων προϊόντων, όχι καταγραφή εκατομμυρίων ενδεχομένω προϊόντων τα οποία απλώ δεν συμμορφώνονται πλήρω με όλε τι απαιτήσει. Και τώρα, όσον αφορά την τελική προσέγγιση, πιστεύω ότι πρέπει να είναι στα χέρια των κρατών μελών. Όσον αφορά τι κυρώσει τώρα, αν και η διατύπωση είναι εν σωστή, νομίζω ότι προβλέπουμε περιβολικά πολλές λεπτομέρειες. Ιδιαίτερα το ποστό κέρδους πρέπει να ληφθεί υπόψη. Άλλο μια εταιρεία με τεράστιο τζίρο και πολύ μικρό περιθώριο κέρδου και άλλο το αντίθετο. Νομίζω ότι το θέμα των κυρώσεων ε, πρέπει να διατυπωθεί με γενικό τρόπο. Αποτρεπτικές και αναλογικέ και να τελειώσουμε εκεί. Και επίση το φόρουμ εποπτεία τη αγορά. Και πάλι εδώ πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Με την ιδέα συμφωνώ εν γέννη. Είναι όμω κάτι το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί σταδιακά από τη βάση μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο των εμπειρογνωμόνων και των άλλων εμπλεκομένων. τέλο, το εργαστήριο αναφορά. Πιστεύω ότι η διάταξη πρόληψη είναι αντιπαραγωγική. Αυτά έχουν γίνει, υπάρχουν το άλλω άλλα εργαστήρια αναφορά σε όλε τι χώρε μέλη. Τα σχολεία μου, λοιπόν, συντείνουν προ καρατούτο ότι είναι μια καλή έκθεση, το λέω και προ τι δύο αλλά νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι και οι και όλοι συνέβαλαν πως ένα καλύτερο κείμενο. Ποιος θέλει να μιλήσει τώρα ή... Α. Άλλος ο οποίος θέλει το λόγο. Ο χρόνος πιέζει. Μπορεί να πάρουμε λίγο χρόνο από τους ε, Σπανού και Βιτόντο. Κυρία Σπανού, ίσως πρώτη. Καλησπέρα κύριε Πιτόντο. Θα μιλήσω και εκ μέρους της κυρίας Μπρίκμαν από την άλλη διευθύνση που δεν είναι εδώ σήμερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω εισηγητές, σκιώδεις. Χαιρόμαστε να ακούμε καλά λόγια τις προτάσεις μας. Ακούσαμε πολλά καλά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά όλα αυτά οφείλονται στο γεγονό, όπως αναγνωρίστηκε ότι Πολλέ από τι προτάσει ε, προέρχονται ούτω ή άλλω από προηγούμενε εκθέσει του Κοινοβουλίου. Άρα πρόκειται για συνεργασία. Κάποια τα οριζόντια θέματα. Καταρχήν, πρόταση για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Ναι, όντω, ο στόχος είναι ένα δίκτυο ασφάλεια. Αυτό ήταν και η αρχική επιδίωξη. Άλλο δίκτυο, άλλο να καλύψουμε τα πάντα. Το λέω αυτό γιατί ο σκοπό μα δεν είναι εδώ θεσπίσουμε νομοθεσία η οποία θα υπερβαίνει την εντολή μας. Θα δούμε τι θα προκύψει από τη συζήτηση, αλλά και πάλι η κεντρική ιδέα είναι ένα δίκτυο ασφάλειας και όχι να καλύψουμε και την τελευταία τρύπα. Η συζήτηση, θυμίζω, έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό επίσης για την προληπτική προσέγγιση υπήρχε μια γενική αρχή η οποία πρέπει να εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Ισχύει είτε περιλαμβάνεται σε ένα κείμενο είτε όχι. Είναι η φιλοσοφία, αν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και δεν περιλαμβάνεται ρητό στο κείμενο. Όχι επειδή την αγνοούμε ή διαφωνούμε μαζί τη. Όχι, ίσα ίσα αναγνωρίζεται ω γενική αρχή η διαφορουμε μαζι τη οχι ισα διέπει όλη την κοινωτική νομοθεσία. έδειξη προέλευση. Το πολλά και προς τις δύο κατευθύνσεις. Να δούμε και εδώ που θα πάει η συζήτηση. Σήμερα ακούσαμε πάντως ότι... Ποιος είναι ο σκοπός εδώ. Ο σκοπός δεν είναι ασφάλεια. Όχι, είναι θέμα ίχνηλασιμότητας. Είναι στο 10% των τριών τα οποία δεν τα βρίσκουμε στο ράπεξ κάθε χρόνο. Μάλλον, συγγνώμη, τα οποία τα βρίσκουμε στο ράπεξ κάθε χρόνο και τα οποία δεν ξέρουμε πού κατασκευάστηκαν, όπου ήρθαν. Θυμίζω για άλλη μια φορά λοιπόν, αν δεν το ξέρετε, ότι πρόκειται για διάταξη η οποία ισχύει στις Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στην Κίνα και είναι και η συνήθις πρακτική. Εδώ απλώ επεκτείνουμε την εφαρμογή της σε προϊόντα στα οποία δεν ισχύει. Για την ένδειξη CE συν το πρόσημο συν. CE τι σημαίνει ότι πληρούν οι απαιτήσει της νομοθεσίας. Ενδιαφέρουσα η πρόταση C+. Επίσης δεν ξέρω αν υπάρχει ανεξάρτητος οργανισμός έγκρισης. Θα το δούμε. Υπενθυμίζω απλώ ότι η ένδειξη CE σημαίνει απλώς ότι ο κατασκευαστής έχει φροντίσει να συμμορφωθεί το προϊόν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ικανοποίηση λοιπόν νομικών απαιτήσεων. Αυτό σημαίνει. αυτό είναι το νόημα του σήματος CE. Όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, διευκρινίζω ότι η πρότασή μας βασίστηκε στην εμπειρία μας από την 358, το 2358, ε, μας αφορά, μας απασχολεί το θέμα του πνιγμού, της ε, κατάποσης, της απόφραξης της θεραπευτικής οδού. Για τέτοιους κινδύνους μιλάμε. Αυτά τα προϊόντα σε αυτήν την περίπτωση υπαγορεύονται. Τώρα άκουσα κάτι για μια διάμεση λύση. Να τα δούμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δεν λέμε όχι. Εξαρτάται από την τελική πρόταση, αλλά θέλουμε μια ισορροπή προσέγγιση, ρεαλιστική και η οποία να συνάδει με την οδηγία. Επίσης σημείωσα αυτό το οποίο είπε η συγγήτρια για την ανάγκη διατλαντικής εργασίας. Ναι, σύμφωνοι, αυτό είναι και το πνεύμα στο Συμβουλίο Γενικών Υπόθεσεων. Μα ενδιαφέρει ο διατλαντικό διάλογο. Ούτω ή άλλω έχω μια ανοιχτή συζήτηση με τι ΗΠΑ. Υπάρχουν εμπόδια, όντω, αλλά σα διαβεβαιώ ότι ω μέλημα παραμένει ε, μέλημα υψηλή προτεραιότητα. Νομίζω ότι κάλυψε τα περισσότερα, αν όχι όλα, όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Πιτικάν. Όντως, στην έκθεση υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Είναι εξαιρετικά ισορροπημένο το κείμενο, επικοδομητικές τροπολογίες. Όσον αφορά τώρα τον κίνδυνο που έχετε από μη συμμορφώσεις, όντως το ακούσαμε και από κράτη-μέλη. Φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη να διευκρινίσουμε τα κινδύνου και της μη συμμόρφωσης. Είναι τομέας στον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε και να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λύση. Η ενημέρωση και η επίγνωση κινδύνου κλπ. Και τα τρία θεσμικά όργανα και τα κρατημέλη νομίζω ότι θέλουν να βελτιώσουν την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς. Όλοι προσπαθούμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Εναρμόνιση όμω κυρώσεων τώρα, πολύ σημαντικό θέμα. Όπω γνωρίζετε η Κομισιόν πρόσφατα πρότεινε ένα καθεστώ για του επισήμους ε, ελέγχου που αφορούν τα τρόφιμα βεβαίω και τι ζωοτροφέ. Είναι κάτι το οποίο ίσω ε, δεν έχει περιέλθει σε γνώσει. Εκεί προτείναμε οι κυρώσει να κυρώνουν ακριβώς το οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο επεδίωξε μια επιχείρηση μέσω της παράβασης. Μπορούμε να εμπνευστούμε από αυτά που γίνονται στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών. Κάτι έχουμε να μάθουμε από εκεί. Τέλο, πολύ σημαντικό, η εξωτερική ανεξάρτητη έλεγχη από τρίτου φορεί είναι μια κοινοφανή προσέγγιση, και καινοτόμος. Δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία. Θα δούμε τι θα προτείνει και το Κοινοβούλιο. Θυμίζω πάντως ότι στο σημερινό σύστημα υπάρχει απέτηση για τεχνική τεκμηρίωση η οποία εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Να δούμε ε, τι στοιχεία έχουμε που μας καλύπτουν από πλευράς ελέγχων και κυρώσεων πριν αλλάξουμε εκβάθρον το σύστημα είναι και θέμα κρατών μελών. Δεν ξέρω αν μπορούν να αντεπεξέλθουν όλα τα κρατημέλη, αν έχουν δηλαδή την δυνατότητα και τι ικανότητε να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα στην πράξη. Ελπίζω να πείτε τα περισσότερα. Για μα έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο ακούσαμε. τηλεφωνική η Λιθουανική Προεδρία μεγάλη σημασία στο να προχωρήσει αυτό ο φάκελο, Θα συνεργαστούμε με τα κρατημέλη και εμεί βεβαίω με το Κοινοβούλιο. Από την πλευρά μα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την λεπτομερή απάντησή σας και σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας, διότι είπα ότι έχουμε του, τις δύο προέδρους, ε, την κυρία Νιμάιστητε, που ασχολείται με την ε, ασφάλεια των προϊόντων των καταναλωτών και τους κύριους Μπαρίσα που ασχολείται με την ασφάλεια των προϊόντων. Εάν θέλετε κάτι να πείτε, μπορείτε ελεύθερα. Απλώς εγώ ανέφερα την παρουσία σας για να, το, για να ξέρουν ότι παρακολουθείτε την εξέλιξη των ζητημάτων αυτών. Λοιπόν, οι εισηγήτριες. Η κυρία Σάλντε Μόζερ και μετά η κυρία Πιέτη Κάινεν και μιλήσουμε και για τα χρονοδιαγράμματά μας. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Δεν νομίζω παρά ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, δεν νομίζω τίποτα άλλο πέραν αυτού. Ας το συζητήσουμε μετά την προθεσμία 4 ε, Σεπτεμβρίου το, στις 12 το μεσημέρι μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Ίσως μερικοί θα πρέπει να εργαστούν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορούμε να εξεύρουμε ε, λύσεις. Δεν μίλησα για την εποπτεία της αγοράς περισσότερο. Ήρθαν σε επαφή μαζί μου πολλοί οικονομικοί φορείς και δεν θέλουν να υπάρχουν νέες προαπαιτήσεις. Μίλησα με πολλά κράτη-μέλη, δεν θέλουν επιπρόσθετο κόστος για την ε, εποπτεία της αγοράς. Κανείς δεν θέλει να επέλθουν αλλαγές, κανένα συμβαλόμενο μέρος, αλλά θα πρέπει να έχουμε ασφαλή προϊόντα στην αγορά και να εργαστούμε προς αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει και οι δύο να υποχωρήσουν και αυτό αφορά και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να φτάσουμε σε μία εξισορροπημένη προσέγγιση. Η κυρία ε, Πίτι Κένεν έχει δίκιο για την εποπτεία της αγοράς, ότι θέλει να την επιτύχει με νέους τρόπους και θα πρέπει να μπορέσουμε να εξεύρουμε νέες λύσεις και να τονίσουμε το ότι οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν πιο ασφαλή προϊόντα στην αγορά και όταν τα σχεδιάζουν και όταν τα ε, θέτουν στην αγορά. Επίσης, ε, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις και σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω την ε, καλή μας συνεργασία κατά τους επερχόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Αυτό αφορά και τους Σκιώδης και την Επιτροπή. Ε, έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την έκθεση, ιδιαίτερα ως προς την πτυχή των κυρώσεων. Και το θέμα της συμμόρφωσης και της αποτίμησης κινδύνων προσβλέπω στην, ε, στους πολύ χρήσιμους συμβιβασμούς και η Επιτροπή και το Συμβούλιο το κατανοούν πλήρως ότι θα πρέπει να κινηθούμε δραστικά. Και αυτό που έχει σημασία είναι να στραφούμε στη σωστή κατεύθυνση για τη νέα αναθεώρηση όποτε και να προβλεφθεί για να δούμε ποια είναι τα μέτρα βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος. Αυτό θα ήταν πολύ ευεργητικό για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και για την ποιότητα των προϊόντων. Προσβλέπω ε, στα σχόλια όλων, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τρόφιμα και ζωοτροφές, μπορούμε πολλά να μάθουμε από αυτές τις προπαρασκευαστικές εργασίες. Δεν θέλουμε να βαρύνουμε ιδιαίτερα τους παραγωγούς κατασκευαστές, ιδιαίτερα όταν ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος όπως το σήμα στη, όχι, στη σωστό, όχι στο σωστό σημείο του προϊόντος. Θα πρέπει να ορίσουμε τους πραγματικούς κινδύνους έτσι ώστε να υπάρξει σωστή κατανόηση στα κράτη-μέλη, ομοιογενής ερμηνεία. Το καλοκαίρι ίσως μας δυσκολεύει τα πράγματα κάπως. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι έγκαιρα θα μπορέσουμε να έχουμε την αποδοχή του κειμένου. Ελπίζω να μας αποστείλετε σχόλια και το Σεπτέμβριο θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, δύο εισηγήτριες εξ ονόματος όλων. Εργαζόμαστε στα πλαίσια ενός ενιαίου πακέτου και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να δείτε την έκθεση εκ του και οι δύο αυτές εκθέσεις αποτελούν παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και βλέπετε ε, τι πιέσει δέχτηκαν από λόμπι, ποιοι είναι οι εμπληκόμενοι φορείς. Αυτό βλέπετε στο τέλος κάθε έκθεσης. Ξέρω ότι πολλοί παρακολουθούν την ανταλλαγή απόψεων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα διαφάνειας και δείχνει και την φύση της εργασίας και συνεργασίας. Ξέρω ότι δέχτηκαν υποδείξεις από όσους ενδιαφέρονται. Απλώς σας επισύρω την προσοχή σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στην ε, κατάληξη, στη λήξη των εργασιών αυτής της Επιτροπής πριν από το ε, καλοκαιρινό διάλειμμα. Έχετε πολλά να επιτελέσετε. Θα ξανασυναντηθούμε στις 5 Σεπτεμβρίου, 5η στις 9 το πρωί. Θα σας δω τότε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Λύεται η συνεδρίαση και θα αρχίσουμε με τους συντονιστές στις 5.30. Sorry. I just want to have the last word uh, uh, of the meeting uh, by thanking Malcolm Harbour being. τον Malcolm Harbour κλείνοντας για την προεδρία του.